Αγαπητές ε, και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί εμπειρογνώμονες εδώ ε, στα έδρανα του προεδρίου, Ας αρχίσουμε λοιπόν, νομίζω και ελπίζω ότι κάποιοι ευρωβουλευτές θα βρουν το δρόμο μέχρι την αίθουσα, όμως αυτό το ότι αρχίζουμε ακριβώς τρεις ορισμένοι το ερμηνεύουν κάπως γενναιόδωρα ας πούμε έτσι. Καλώς ήρθατε στην σημερινή συνεδρίαση με τον τίτλο Scientific Culture Αντίδραση στις ψευδείς ειδήσει. Το πρόβλημα που ε, κρύβεται από πίσω είναι η πολιτική ριζοσπαστικοποίηση από τις μεγαλύτερες και δυνότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Τώρα και μετά από το δημοψήφισμα για τη Βρετανική αποχώρηση και τις εκλογές του νέου Αμερικανού Πρόεδρου έχει γίνει ακόμα πιο ε, καυτό το θέμα αυτό και στο διεθνές αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο χρησιμοποιούνται οι ψευδείς ειδήσει για χειραγώγηση των πολιτών και της κοινή γνώμης με τελική ε, επίπτωση υπονόμευση της δημοκρατικής τάξης. Ιδίως για τη δική μας επιτροπή που ασχολείται με την εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να κηρύξει τον αγώνα κατά των fake news και των εναλλακτικών αληθιών όπως τα λένε εφημιστικά που δεν είναι παραψέματα. Γι' αυτό και χαίρομαι που έχουμε κοντά μας σήμερα πέντε διεθνείς εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα μας φωτίσουν διάφορες πτυχές του θέματος και ιδίως το ερώτημα σχετικά με τις δυνατότητες αντιμετώπισης με επιστημονικό τρόπο των ψευδών ειδήσεων. Η ακρόαση χωρίζεται σε δύο μέρη. Και μετά από κάθε γύρο θα ακολουθεί γύρος ερωτήσεων και απαντήσεων, ώστε να έχουμε επαρκή χρόνο για να αναπτυχθεί μια συζήτηση. Το πρώτο πάνελ περιλαμβάνει τους εξής ε, τρεις διεθνούς εμπειρογνώμονες, Νικολάη Ναϊντένοφ, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Σόφια που θα μιλήσει για την cryptical approach στην πολιτική των fake news. Ακολουθεί ο κύριος Vincent Χέντριξ καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης, ο οποίος θα μιλήσει για fake news και κοινωνική ψυχολογία. Και ο Μάσιμο Μαρκιόρη, Μάσιμο Μαρκιόρη, καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάδουα, ο οποίος θα μιλήσει για μηχανές αναζήτησης και χειραγώγηση της αλήθειας. Καλώς ήρθατε λοιπόν και οι τρεις εδώ στην Επιτροπή μας και σας υπενθυμίζω ευθύς αμέσως ότι οι παρουσιάσεις σας ε, θα πρέπει να αρκεστούν σε 10 λεπτά για να δοθεί χρόνος και για συζήτηση. Θα βάλω μπροστά το χρονόμετρο και θα σας κάνω ένα ήπιο νεύμα εάν υπερβείτε τον χρόνο σας για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα να δώσω τον λόγο στον κύριο Ναϊντενόφ για 10 λεπτά. Ορίστε κύριε, έχετε τον λόγο. Dear Mrs. dear members of the European Parliament. Ε, αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, ε, μέλη της Γραμματείας, είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να συζητήσω κάποια καυτά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σύγχρονης δημοκρατίας. Τα... Θα μιλήσουμε για τα fake news και πώς αυτά χαρακτηρίζονται. Πρώτη διαφάνεια. τον τίτλο. Μιλάω για κοινική προσέγγιση, γιατί υπάρχει μια αντίφαση. Από τη μια αποφεύγονται οι δημοκρατικοί μηχανισμοί με τα fake news και επιδιώκονται πολιτικά αποτελέσματα, επικαλούμενοι, ε, κοινωνικό στάτους, ε, εθνικές ιδιαιτερότητες κλπ. Από την άλλη, ε, στη, ε, προσπαθούν να αλλάξουν την συμπεριφορά των ανθρώπων. These two lessons Και να επηρεάσουν τις εκλογές. Εδώ βλέπετε τις πιο συντριπτικές ε, ε, επιπτώσεις των fake news που αποτελούν και την καρδιά του σύγχρονου υβριδικού πολέμου. Οι στόχοι είναι πάρα πολλοί, αλλά οι πολιτικές χρήσεις είναι τρεις. Εγώ θα αναφερθώ στο τρίτο που αυτό σημαίνει ότι η αξιολόγηση του τι είναι ψεύτικο στις ειδήσει ε, απαιτεί μία μελέτη ε, της γενικότερης ροής των ειδήσεων. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε πώς ερμηνεύονται στα πλαίσια του υβριδικού πολέμου τα fake news. Ε, χρησιμοποιούν εσωτερικές ε, σχέσεις και ο κινησμός ε, δημιουργεί και ο ίδιος ειδήσει. Ε, βλέπουμε ε, την εξάπλωση ε, των fake news και πώς επηρεάζουν κοινωνικά φαινόμενα και πώς έχουν και εξωτερική επιρροή. Τα fake news ε, προσπαθούν να εμβαθύνουν, να βαθύνουν τη διαφορά μεταξύ πολιτικών ελίτ και εκλογικού σώματος. Επίσης, ε, χρησιμοποιούν μηχανισμούς ε, που, τους κάνουν, που τα κάνουν δυσδιάκριτα από τους ερευνητές. Έτσι είναι δύσκολο να καταδειχθούν έχω αναφέρει κάτι σημαντικό επίσης, ότι τα κατάλοιπα της κομμουνιστικής προπαγάνδας είναι ε, το καλύτερο έδαφος για την εξάπλωση των fake news. Υπάρχουν τρεις τρόποι για τη διάδοση των fake news. Κυρίως όμως πολλαπλασιάζονται τα fake news από τον ίδιο τον κόσμο με προσωπική επικοινωνία, με τα κοινωνικά μέσα. Ε, έτσι ξεφεύγουν και από το δημόσιο έλεγχο, χειραγωγώντας ε, απόψεις ε, και χειραγωγώντας και τις αντιδράσεις στις εξελίξεις των ανθρώπων. Τα fake news διαδίδονται και από χώρες και από οργανισμούς, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι οι χώρες που διαδίδουν τα fake news. Χώρες με αντιφατικό προφίλ. Από τη μια δεν είναι αρκετά πλούσιες για να έχουν πολιτική επιρροή που θα ήθελαν να έχουν, αλλά έχουν πόρους ε, φυσικούς Μεθοδολογικά τα fake news στηρίζονται στα κατάλοιπα των ε, παλιών παραδόσεων της κομμουνιστικής προπαγάνδας. Αυτές οι παραδόσεις έχουν ηλικία 100 ετών. Τώρα πια. Και φτάνω σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και θα αναφέρω ε, κάτι ασυνήθιστο. Κάποιες αντιφατικές τάσεις δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια καταστρέφουν ή παραλύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, αν θέλετε, σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο ενάντια στα fake news. Γι' αυτό έχω συμπεριλάβει και αυτά τα σημεία. Ποιες είναι αυτές οι τάσεις. Εδώ ε, εντοπίζω κάποιους τομείς και τάσεις. Υπάρχει, για παράδειγμα, ε, μια διαφορά μεταξύ δημοσίου χώρου, ιδιωτικού χώρου, δημόσιο αφήγημα, ιδιωτική ζωή, ε, την κοσμικεύση του κράτους, την, το διαχωρισμό εκκλησίας κράτους, τα ταμπού, Ε, πολλές φορές ε, ακόμα και οι κοινωνικές επιστήμες ε, γίνονται πολύ εμπειρικές έτσι αφήνουν ή παραμελούν το θεωρητικό κομμάτι. Αυτά όλα οδηγούν σε μείωση της ζωτικότητας της κοινωνίας. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Πρέπει να σταματήσουμε την αρχιετυπική κοινωνική διάκριση ε, για να ε, αντιμετωπίσουμε διαφορές και ανισότητες. Ε, πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την ισότητα μεταξύ των φύλων με τις διαφορετικές παραδόσεις ε, άλλων πολιτισμών, πώς ε, επηρεάζονται τα media arts και η ζωητικότητα της ίδιας της κοινωνίας. Για παράδειγμα, ε, το, η παράδοση του ουμανιστικού κινηματογράφου έχει εξαφανιστεί. διαφοροποιούνται και τα προγράμματα στην τηλεόραση και βλέπουμε πολύ ε, ε, μεγάλη επιδίνωση της ε, ποιότητας. η ανεκτικότητα έχει υποβαθμιστεί. Επίσης υπάρχει προβολή των διαφορετικών χαρακτηριστικών έναντι των άλλων ε, πολλές φορές μπαίνουν σε κουτάκια οι άνθρωποι ανάλογα με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, θρησκεία κλπ. Αν τονίζονται μόνο οι διαφορές μεταξύ πολιτισμών, δεν αναγνωρίζουμε τις ομοιότητες και τα κοινά σημεία. Τα ε, προβλήματα λοιπόν αυτά μπορούν να λυθούν ε, μόνο όταν υπάρξει ε, μια ε, πιο ρωμαλαία κοινωνία η οποία θα μπορέσει να συγκεράσει τις διαφορετικότητες. Χρειάζεται επίσης και χρειάζονται μέτρα διοικητικά, μέτρα που θα ληφθούν από τον δημόσιο τομέα. Final effects. Such trends which endanger the ε, όλα αυτά οδηγούν σε πολιτική διαφθορά και αποτελούν εσωτερική και εξωτερική απειλή για την Ένωση. Αυτό δεν το είχα αναφέρει στις διαφάνειες. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρωσε μεγάλο τίμημα από τα προβλήματα που προέκυψαν από το Brexit, τις αυτονομιστικές τάσεις στην Καταλωνία κλπ. Η αντίληψή μου για τα fake news ε, που βρίσκονται ε, ε, στην καρδιά του υβριδικού πολέμου είναι αντικείμενο πολιτικών, των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών και όχι μόνο. Εδώ παρουσιάζω μια σκέψη του Άντλαϊ Στίβενσον στο τέλος. Και συμφωνώ όταν λέει ας ε, ε, προσπαθήσουμε να πείσουμε ε, και να καταδείξουμε τη λογική στον Αμερικανικό λαό. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος, τον Ευρωπαϊκό λαό δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ για, τις, για τα εισαγωγικά σας λόγια. Ο κύριος Χέντριξ λαμβάνει το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Θα μιλήσω για το φιλόξενο περιβάλλον για τα fake news από την κοινωνιολογική άποψη και τους σχετικούς μηχανισμούς. Ας ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα πρώτα και ας δούμε την αγορά πληροφορίας ή την ψηφιακή εποχή ως αγορά ψηφοφορίας. Ένα χαρακτηριστικό έχει και το αντιλαμβανόμαστε ήδη. Ο Σάιμαν από το 1979 μας είχε πει ότι βασικά αυτό που προσπαθείς να αποσπάσεις είναι η προσοχή των άλλων ανθρώπων και έτσι καταναλώνονται οι πληροφορίες. Αυτά βέβαια έχουν και ένα τίμημα. Εάν κατανοήσει κανείς ένα πράγμα ότι το βασικό δηλαδή είναι η προσέλκυση της προσοχής θα υπήρχε μια δημοκρατική έννοια της κατανομής της προσοχής αν δινόταν δηλαδή η προσοχή σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες. Όμως η προσοχή δεν κατανέμεται. Δεν σημαίνει ότι όλοι από εμά λαμβάνουμε ίσο μερίδιο προσοχής από άλλους ανθρώπους. Αλλά εκεί ισχύουν οι νόμοι της δύναμης, της εξουσίας. Υπάρχουν ορισμένε ομάδες, είτε μιλούμε για μεγάλες ε, μεγάλους φορείς που προωθούν πληροφορίες στο διαδίκτυο κλπ. Αυτοί προσελκύουν την προσοχή των πολλών και οι υπόλοιποι αναγκάζονται να αγωνιστούν για να αποσπάσουν την προσοχή των ολίγων. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Εάν επιστρέψουμε στον φονταμενταλισμό της αγοράς από την αρχή του, 2000, είχαν πει τότε ότι η ελευθερία στην αγορά θα εξασφαλίσει την ισορροπία και ότι οι καλής ποιότητας υπηρεσίες θα κατησχίσουν και οι υπόλοιποι θα εξαφανιστούν. Ακόμα και όλαν Greenspan τα έλεγε αυτά. Όμως αυτά κατέληξαν στην κρίση του 2008 και κατέληξαν, εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα ότι οι χρηματοοικονομικές αγορές και υπηρεσίες δεν λύνουν το πρόβλημα, παρόλο βεβαίως που οδήγησαν σε κακά πιστοτικά προϊόντα. Εν τέλει, οι ψεύτικες ειδήσει είναι ένα κακό προϊόν και επειδή δεν είναι αποτελεσματική αγορά και όλοι οι λόγοι συνηγορούν υπέρ αυτής της απόψεως, ας αντιληφθούμε ένα πράγμα. Κάθε χρήστη κοινωνικών μέσων όπου κυκλοφορούν και πολλαπλασιάζονται ειδήσει αληθινέ, ψεύτικες, bullshit που λένε στα αμερικάνικα, δηλαδή αειδίε, αρκεί να κατανοήσουμε όλοι ότι εμεί είμαστε οι πελάτε του Facebook ή τουλάχιστον οι χρήστε. Αλλά α θεωρήσουμε αυτού ω πελάτε των κοινωνικών μέσων Ακόμη και έτσι ε, δεν έχουμε κατανοήσει σωστά το μοντέλο με το οποίο τα κοινωνικά μέσα βγάζουν λεφτά. Ως εξή λειτουργούν. Οι χρήστε πρέπει να προσφέρουν κάποιες πληροφορίες, τις οποίες πληροφορίες τις χρησιμοποιούν άλλοι χρήστες. Τις κάνετε μια δέσμη πληροφορίες αυτές και τις πουλάτε σε άλλους. Ποιους? Στους διαφημιστές. Και αυτό είναι το προϊόν. Τονίζω ότι μόνο και μόνο επειδή είμαστε χρήστες δεν είμαστε πελάτες. Είμαστε το προϊόν στην πραγματικότητα εμείς οι χρήστες. Και είναι τελικώς η happy hour για τις ψευτείς ειδήσει. Μπορεί να υπάρξει μια εισβολή ψευδών ειδήσεων, αυτό έτσι το λέμε. Και αυτό έχει σχέση με τον τρόπο που έχει δημιουργηθεί αυτή η αγορά των πληροφοριών. Πώς έφτασαμε εκεί, υπάρχει ένας ορισμός των fake news. Εύκολα μπορεί να το πει κανείς Α υποθέσουμε ότι υπάρχει μια αλήθεια και υπάρχει κάτι που είναι ψεύδο. Άλλε φορέ είναι εύκολο να διαπιστωθεί αλήθεια, άλλε φορέ δύσκολο. Τουλάχιστον α αντιληφθούμε ότι υπάρχει μια διάκριση μεταξύ αλήθεια και ψεύδου που πρέπει να το αντιληφθούμε. Ακόμα και οι ψεύτε αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ αλήθεια και ψεύδου. Αλλιώ δεν ξέραν οι ίδιοι ότι είναι ψεύτε. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο ψεύτη είναι τουλάχιστον ειλικρινή κατά την έννοια ότι αντιλαμβάνεται ότι αυτό που λέει είναι ψεύδο. Όμως αυτός που χρησιμοποιεί BS, bullshit δηλαδή, ideas, δεν δέχεται την διάκριση μεταξύ αληθούς και ψευδούς. Αυτό το έχει εξηγήσει ο Χάρη Φράνκφορτ σε ένα μικρό βιβλίο που το λέει on BS, bullshit δηλαδή. Δεν, το λέει, δεν λέει τη λέξη ολόκληρη δηλαδή. Αυτό που λέει με λίγα λόγια είναι το εξής. Αυτός που χρησιμοποιεί το bullshit, τις αηδίες, δεν δέχεται την διάκριση μεταξύ αληθού και ψευδού. Μπορεί να τα ανακατέψει αυτά όπω θέλει. Να πάρει λίγα αληθινά πράγματα, λίγα ψεύτικα πράγματα, με διαφορετικού σκοπού κάθε φορά. Και συνήθω αποκρύπτει τα κίνητρά του. Μπορεί να είναι προπαγάνδα, μπορεί να είναι για λεφτά ή μπορεί να είναι για τρολάρισμα. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικά κίνητρα για την παραγωγή των ψευδών ειδήσεων, αλλά υπάρχει όμως και χρηματοδοτικό κίνητρο, διότι κάνει φασαρία, είναι εντυπωσιακό και παράγει χρήμα. Κάθε τι που είναι αλήθεια δεν σημαίνει ότι είναι και viral, ότι διαδίδεται γρήγορα στο διαδίκτυο. Ούτε και το αντίθετο. Αυτό έχει αποδειχτεί τα τελευταία δέκα χρόνια κατά επανάληψη. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικά είδη ποιότητα τη πληροφορία. Α δούμε ένα είδο κλίμακα. Στην πρώτη ζώνη έχετε αλήθεί ειδήσει. Μετά έχετε τα άλλα τα οποία τα έχουν πειράξει, doctor statements. Δεν είναι απαραίτητα λάθη, αλλά τα βάζουν σε κάποιο πλαίσιο και με πολλού, πολλούς τρόπους μπορείτε να πειράξετε, να διορθώσετε κάποιες αληθείς πληροφορίες ανάλογα με το τι θέλετε, πώς θέλετε να προσελκύσετε την προσοχή των ανθρώπων αφού κάνετε προσεκτική επιλογή των όσων θέλετε. Τι θέλετε, 10% ανεργία ή 90% απασχόληση. Έχει διαφορά, παρόλο που το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν μετά σε τρίτη κατηγορία ζώνη 3 τα ψέματα. Τα ψέματα είναι ψευδή. Όμως επίτηδες παρουσιάζονται ότι έρχονται σε αντίφαση με οτιδήποτε είναι αληθές. Και μετά, όπως σας είπα, έρχονται και το bullshit, το οποίο πλέον έχει γίνει αποδεκτό σε επιστημονική ορολογία και ε, τίνει να δείξει την, την κατάργηση των διακρίσεων μεταξύ αληθούς και ψευδούς. Και αυτό είναι εν τέλει η ψευδής είδηση. Η ψευδής είδηση είναι μια δήλωση bullshit η οποία εμφανίζεται σαν δίθεν αληθής και σαν δίθεν δημοσιογραφία ενώ δεν είναι. Και αυτό είναι που την κάνει δηλητηριώδη διότι όταν δεν αποδέχεστε τη διάκριση μεταξύ αληθούς και ψευδούς μπορείτε να πείτε οτιδήποτε θέλετε αρκεί να κάνετε φασαρία με τον τρόπο αυτό. Και η φασαρία έχει σημασία εδώ διότι υπάρχουν μελέτες που δείχνουν με ξεκάθαρο, κρυστάλλινο τρόπο από το Πανεπιστήμιο της ε, Κολάμπια. Δείχνουν λοιπόν ότι ένα κλειστό οικοσύστημα στις, στις ε, αμερικανικές εκλογές του περίφημης, της περίφημης του σελίδας Brightband μπόρεσε να δημιουργήσει ένα κλειστό οικοσύστημα όπου μιλούσαν σε ένα συγκεκριμένο είδος ανθρώπων στους οποίους ήθελαν να απευθυνθούν στους λευκούς Αμερικανούς ας πούμε ένα, μια ειδική δημογραφική ενότητα και θέλαν να τους πούνε πράγματα που αυτοί θέλαν να ακούσουν κάνοντάς το με τέτοιο τρόπο εντυπωσιακό ώστε αναγκάστηκαν να τους προσέξουν τα υπόλοιπα, τα ε, συστήματα παροχής πληροφοριών, τα υπόλοιπες εφημερίδες κλπ δεν υπάρχει καλή ή κακή προσοχή. Είτε έχετε την προσοχή του κοινού είτε όχι. Και αυτό που σας απασχολεί να προσελκύσετε την ε, προσοχή. Και το fake news έχει κάποια αξία. Δηλαδή, αν θέλουμε να έχουμε στοιχεία για να λάβουμε μια απόφαση, τι κάνουμε. Κοιτάμε τι κάνουν οι άνθρωποι γύρω μας. Οκ, βλέπετε και την καρικατούρα. Και στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης έχουν κάνει τις λεγόμενες bubble studies, μελέτες της φούσκας που δημιουργείται και δείχνει ότι υπάρχουν ψυχολογικοί μηχανισμοί από πίσω. Και είναι αλήθεια το γεγονός ότι πάντοτε είμαστε ευαίσθητοι στην επιρροή των άλλων. Ποτέ δεν έχει αλλάξει αυτό, ούτε βεβαίω στην εποχή της πληροφορικής. Αντίθετα, έχει γίνει πιο δυνατή αυτή η επιρροή. Είναι αυτό το bystander effect. Δηλαδή, ακούμε τι λέει ο διπλανός μας και επηρεαζόμαστε και υπάρχουν πάρα πολλέ ε, ορολογίες κυρίως αμερικανικής εμνεύσεως που λειτουργούν μια χαρά στην ε, εποχή της πληροφορικής. Και μετά χρησιμοποιήστε fake news για να τους κάνετε όλους να κοιτάξουν προς την ίδια κατεύθυνση. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ε, επιχειρηματολογία σχετικά και δημιουργείται μια απολύτως νέα κατάσταση που γίνεται αποδεκτό να χρησιμοποιηθούν αυτά που λέμε blue lies, τα κιανά ψέματα. Δηλαδή ψέματα που τα λέει κανείς για λογαριασμό της ομάδας και αυτό τα κάνει αποδεκτά και αυτό που οδηγεί στην πόλωση σε ένα είδος ε, ταυτότητας φυλής, ταυτότητας ομάδας μέχρι ενο σημείου όπου αυτοί που ανήκουν στην ομάδα, στη φυλή είναι πλέον ανθεκτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε επιρροή απ' έξω. Θυμηθείτε την φωτογραφία το, της ανάληψης καθηκόντων του Ομπάμα και του ε, Τραμπ και την τεράστια διαφορά τα πλήθους. 40% των ε, οπαδών του Τραμπ θεώρησαν ότι όντως παρόλη τη φωτογραφία ήταν περισσότερος ο κόσμος που είχε πάει για τον Τραμπ. Τόσο τέτοια μπορεί να είναι η πόλωση όταν η πόλωση αυτή είναι αρκετά μαζικού χαρακτήρα. Και μπορείτε να το δείτε τα fake news σαν ένα πραγματικό όχημα για την επιβολή ατυχών παγίδων όπου μπορεί να το, μπορείτε να κάνετε το κοινό να πέσει μέσα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Η πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ, πραγματικά πολύ. Θα ακολουθήσει ο κύριος Μαρκιόρη. Έχετε το λόγο κύριε για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ που ε, με ε, καλέσατε εδώ. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Πολλά πράγματα ε, μπορούμε να πούμε όσον αφορά το θέμα αυτό θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι ενδεχομένως μόνο τα κοινωνικά δίκτυα είναι η τεράστια πηγή από την οποία αντλούμε τα fake news. Όχι, αυτό δεν ισχύει όμως. Είναι πολλοί αυτοί οι παίκτες οι οποίοι παίζουν ε, σημαντικό ρόλο. Η πληροφορία βεβαίως και η πληροφόρηση παίζει ε, σημαντικό ε, ρόλο αλλά εξαρτάται και από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται και κατανοούν τις μηχανές αναζήτησης οι χρήστες ε, και συμπληρώνονται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ε, ε, και αλληλοεπιδρούν τα κοινωνικά μέσα με τις μηχανές αναζήτησης. Είναι σημαντικό ε, ε, κάτι ε, αξίζει τον κόπο να αγωνιστεί κανείς γι' αυτό. Εάν θέλεις να προσπαθήσεις να πείσεις τους άλλους θα πρέπει να πάρεις την πρώτη θέση και εάν δεν πείσεις με την πρώτη ματιά τότε το ένα περίπου 50% φεύγει από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή το 50% του 51% 3%, συγγνώμη, τα 3% τέταρτα των ε, ακροατών ε, και εάν κάνεις το ίδιο πράγμα μια δεύτερη φορά τότε μπορεί να χάσεις μέχρι και 93% και, ε, και δεν υφίστασε, δεν υπάρχει εάν δεν είσαι στους 10 πρώτους που θα βγουν από την μηχανή αναζήτησης και δεν πρέπει να μας εκπλήσει η μεγάλη διασύνδεση που έχουν οι μηχανές αναζήτησης και τα αποτελέσματά τους με τα κοινωνικά δίκτυα, αυτά τα δίκτυα κοινωνικά κοινωνικής όπως τα λέμε. Ε, ε, όταν κάτι επαναλαμβάνεται και ξανά ε, αναφέρεται τότε η ορατότητα είναι πολύ μεγάλη. Γίνεται αυτό που ονομάζουμε αντίχηση. Βεβαίως ο κόσμος... προσπαθεί να βρει κάτι ε, στο Google ας πούμε και τα πρώτα 10 αποτελέσματα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που ε, έχει ε, ψάξει γιατί ενώ ψάχνει για τον Λόρδο Βύρονα μπορεί να του βγει κάτι οτιδήποτε άσχετο το οποίο όμως έχει μέσα τη, λέξη Βύρον και επομένως καταλαβαίνετε ότι με τον τρόπο αυτό είναι απολύτως θρευλή η εικόνα και η πληροφόρηση που έχει. Ε, υπάρχει επίσης και μια χρονική διαστρωμάτωση. Ε, ε, κανείς μπορεί να σκεφτεί ότι τα fake news δεν είναι ακριβώς λάθος ψεύτικη πληροφόρηση. Όντως είναι ένα πολύ γενικότερο φαινόμενο το οποίο αφορά την πληροφόρηση αλλά χρησιμοποιεί και την, αυτήν την χρονική ας πούμε ε, αλληλουχία ε, και ε, με τον τρόπο αυτό μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα με πιο αργό ρυθμό και επομένως να μην μπορέσουν να εσωματωθούν οι αλλαγές. Μπορεί να γίνουν οι αλλαγές με πολύ χαμηλότερο, πολύ πιο χαμηλό ρυθμό και ταχύτητα αλλά παρόλα αυτά το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μονάχα τα fake news αλλά όλα τα ε, μέσα. Ένα πολύ καθαρό παράδειγμα είναι η Wikipedia. Είναι η εγκυκλοπαίδεια των ε, δικών μας ε, χρόνων, της δικιάς μας εποχή είναι ένας πρωτογενής ε, στόχος ε, αυτή η ε, Wikipedia. Η Wikipedia βγαίνει πάντα στις τρεις πρώτες, στα τρία πρώτα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης Google. Και λένε ότι η Wikipedia μπορεί να, έχει, μπορεί να κάνει επίτηδες κοινωνικό έλεγχο. Ε, δεν είναι ακριβώς έτσι, ε, αλλά μέσα από την παρίσφρηση ψευδών στοιχείων μπορεί κανείς σιγά σιγά και με τη διαδικασία που ανέφερα προηγουμένως να αλλάξει ακόμα και ιστορικά γεγονότα. Έχουμε επίσης ε, τώρα και την ε, Negapedia, βγαίνει από το Google. Ε, είναι μια αρνητική εκδοχή της Wikipedia και και βλέπεις ότι πίσω από κάθε ε, σελίδα υπάρχει και το κατά κάποιο τρόπο υποπροϊόν αυτής της ε, σελίδας ε, όπου αναφέρεται μία άλλη άποψη, ενδεχομένως το fake news το οποίο κρύβεται εκεί. Πάντως πίσω από αυτά που βλέπουμε σαν πρώτη πληροφόρηση από τη Wikipedia μπορεί να κρύβονται πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι γραμμική εντωμεταξύ η οδός που ακολουθούν αυτές οι ε, διαδικασίες. Ε, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν κάποια κατόφλια αλλά μπορεί να προκύψουν και οι λεγόμενες χιονοστιβάδες, δηλαδή κάποιες ε, καταστροφές, ένα είδος cascade effect. ο κοινωνικός μας, ε, ο, ο, κόσμος μας πλέον είναι υπερσυνδεδεμένος ε, και η δύναμη του αντλείται ακριβώς από αυτήν την υπερσύνδεση γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε, είναι ο τρόπος με τον οποίο πληροφορούμαστε ε, και εδώ ακριβώς ξεκινάει η, η δυσκολία. Φυσικά υπάρχουν και κάποια καλά νέα με την έννοια ότι είναι αρκετά εύκολο να ξεκινήσει κανείς ε, ε, να φτάσει μέχρι το ε, κατόφλι αλλά όταν περάσει το πρώτο κατόφλι ε, τότε μπορεί η κατάσταση να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνη. Προς τα πού πηγαίνουμε μπορεί να αναρωτηθεί κανείς. Ε? Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς την εξελικτική ανάλυση, μπορεί να χρησιμοποιήσει μοντέλα, τη μοντελοποίηση δηλαδή για να δει πού μπορούμε να οδηγηθούμε. Μπορεί να κάνει και αυτό τον, να βρει και τον συσχετισμό ανάμεσα στο όφελος και την ε, ζημία. Ε, αλλά εάν κανείς είναι προσεκτικός θα καταλάβει ότι αυτός ο συσχετισμός ωφέλους ε, και ζημίας είναι πάρα πολύ αρνητικός για μας. Τι λύση μπορούμε να βρούμε. Πρώτα απ' όλα να δώσουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια του περιεχομένου έτσι ώστε να μην είναι το κυριότερο, η πρώτη προτεραιότητα το να βάλει κανείς το ψεύτικο περιεχόμενο, να είναι σαφές ότι αυτό είναι ε, ε, κακό. Θα πρέπει οπωσδήποτε να πιέσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, ε, γιατί είναι σημαντικό να δώσουμε μεγάλη σημασία στην ίδια την πληροφόρηση στην αρχή, γιατί μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεύτερος, δεύτερος, κανόνας είναι η διαφάνεια ε, ε, ε, λέμε ναι είναι αυτοί οι οποίοι κρατάνε τα κλειδιά του βασιλείου της πληροφόρησης αυτές οι μηχανές. Ναι αλλά και εμείς είναι ανόητο να το πούμε αυτό αν το σκεφτεί κανείς γιατί εμείς βάζουμε τα στοιχεία αυτά. Όλοι μας λένε ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ναι αλλά δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια μέσα από, την, το σκοτεινό ίντερνετ. Θα πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να προστατευτούμε. Και υπάρχει μια λύση. Είναι η, η, η βιώσιμη μορφή ε, α, διαφάνειας. Ε, μια διαφάνεια δηλαδή βάσει της οποίας εμείς ε, σαν κοινωνία θα μπορούμε να ελέγχουμε ακριβώς το τι συμβαίνει με τις πλατφόρμες και τι συμβαίνει με την κατάσταση αυτή. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως αυτό ακριβώς να αποτελεί ε, και την κρυφή συνταγή για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε ε, τα προβλήματα. Μπορούμε λοιπόν να πάμε να ελέγξουμε, να δούμε ε, ε, σε άλλες μορφές της ε, κοινωνίας μας, να πάμε να δούμε πώς κάνει τη δουλειά της η coca ή τι γίνεται σε μια άλλη διαδικασία. Το ίδιο θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε και με την πληροφόρηση. Δηλαδή διαφάνεια και σωστή πληροφόρηση, γιατί η πληροφορία ακριβώς είναι η τροφή του μυαλού μας και δεν μπορεί να είναι δηλητηριασμένη η τροφή αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος Κάμερ Εύερτ. Πολύ ενδιαφέρουσες οι προτάσεις, οι ιδέες που ελπίζω ότι θα προκαλέσουν και ερωτήσεις και συζήτηση στην, ε, στον επικείμενο γύρο. Αν συμφωνείτε, θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στους συντονιστές μας και μετά στα υπόλοιπα μέλη αναλόγως με την σειρά που θα ζητήσουν το λόγο. Πρώτη, κυρία Σαμπίνε Φερχάιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για όλες τις ε, παρουσιάσεις που και για μας ε, είναι πολύ διαφωτιστικές. Δύο θέματα. Πώς αναλύω τα fake news και πώς συμβαδίζουν οι αναλύσεις αυτές με τις δημοσκοπήσεις και τις ε, δημοσιογραφικές έρευνες. Συνήθως στα κλασικά μέσα ενημέρωσης έχω το λεγόμενο impressum, δηλαδή γνωρίζω ποιος υπογράφει. Στο διαδίκτυο αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν και ιδίω στα ε, διάφορα δίκτυα, κοινωνικά δίκτυα και άλλα, δεν υπάρχει καμιά επαλήθευση και ηθελημένα δεν υπάρχει. Πώς λοιπόν μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. Δεύτερο, η αντίχηση, για παράδειγμα, υπάρχει στα ε, κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή παρακολουθώ και ε, επιβραβεύω με το like μου πράγματα τα οποία μου αρέσουν και αυτά πολλαπλασιάζονται. Ενώ υπάρχει τάση από αυτή την αυτοαντιλαμβανόμενη αλήθεια δεν αντιλαμβάνομαι πλέον τι είναι αληθές και τι είναι ψεύδος διότι θεωρώ ότι η αλήθεια που μου παρουσιάζει τη αλήθεια είναι αλήθεια και επομένω τελικώ συγχαίεται με την πραγματική αλήθεια και χάνονται τα γεγονότα. Πώ μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Τρίτο, οι μηχανέ αναζήτηση, τι οποίε δείξατε προ το τέλο τη ε, ε, ε παρουσιάσεώ σα και που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Πώς μπορεί ενδεχομένως να γίνει κάποια ρύθμιση εκεί και μπορεί να είναι στόχος μας Ούτω ή άλλω, το Google στη βάση των αλγορίθμων που χρησιμοποιεί κάνει κάποιε επιλογέ. Και ω Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθήσαμε κατά επανάληψη να προσεγγίσουμε αυτού του αλγορίθμού και να δούμε εάν μέσω των αλγορίθμων οδηγούμαστε και σε στρέβλωση του ανταγωνισμού στι αγορέ, Έχουν μάλιστα επιβληθεί και χρηματικέ ποινέ, πρόστιμα δηλαδή στο Google και τώρα μάλιστα ε, πρόκειται να επιβληθεί. Πώ μπορεί να τα ρυθμίσει κανείς αυτά. Πρέπει να τα ρυθμίσει κανεί αυτά, νομοθετικά εννοείται. Πώς, εσύ είναι οι αντιλήψεις, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε εκτός από την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, των πολιτών, αμφωτέρων των φίλων εννοείται, και ότι να αντιληφθούν ότι δεν είναι πάντοτε αλήθεια αυτά που βλέπουν στο διαδίκτυο. κυρία Κώστα, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ε, όλους τους παρεμβαίνοντες ε, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσατε ε, τα διάφορα θέματα και ευχαριστούμε και για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε. Αυτό το θέμα των μηχανών αναζήτησης μας απασχολεί πάρα πολύ και θα πρέπει να δούμε και το θέμα των αλγορίθμων και τον τρόπο με τον οποίο Όλη αυτή η προβληματική συνδέεται και με τα κοινωνικά δίκτυα. Το ζήτημα είναι όμως να μπορέσουμε και με τη, σε συνεργασία με τις πολιτικές ε, ε, αρχές, σε εθνικό, διεθνές επίπεδο, ε, να απαιτήσουμε ε, κάποιες ε, διαφαν... κάποιους διαφανείς κανόνες, κάποια αντικειμενικότητα από τις μηχανές αναζήτησης, γιατί το θέμα των αλγορίθμων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, θα ήθελα να ξέρω άν κατά την άποψή σας υπάρχει βέβαια από τη μία μεριά η δυνατότητα να ενισχυθεί η κριτική σκέψη, αλλά αυτό είναι ένα θέμα γενικότερη της εκπαίδευσης ε, το οποίο δεν αρκεί. Εμείς ε, θεωρούμε ότι οι πλατφόρμες οι οποίες δεν είναι μόνο hosting αλλά είναι ε, proactive θα πρέπει να ελέγχονται. Όσον αφορά τα κοινωνικά δίκτυα το θέμα είναι πιο περίπλοκο. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ή ορισμοί. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια έτσι ώστε να βρούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να απαγορεύσουμε τις εσκεμμένες ε, εκστρατείες επιρροής της γνώμης πως είναι δυνατόν ε, αυτό το ίδιο σώμα το οποίο αναφέρατε προηγουμένως ε, να παράγει τα δικά του αντισώματα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει και αντίκτυπος όχι μονάχα στην δημοκρατία, όχι μονάχα σε σχέση με την, με την, ε, με την ε, διαφάνεια κτλ. Αλλά υπάρχει στην ουσία οπισθοδρόμηση, ε, μια επιστροφή σε παλαιότερα μοντέλα τα οποία μπορεί να έχει πολύ κακές επιπτώσεις ακόμα και για θέματα τα οποία αποτελούν πεδίο επιστημονικό. Βλέπουμε ε, ότι λόγω ακριβώς ε, της ε, ψεύτικης, των ψεύτικων επιστημονικών δίθεν ειδήσεων έχουμε μία μείωση ας πούμε των εμβολιασμών που φτάνει και ξεπερνάει το 30%. Αυτή λοιπόν είναι μία κακή πληροφόρηση, μία αντίθετη πληροφόρηση η οποία πίσω από μανδύα επιστημονικό κάνει πάρα πολύ κακό. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τα ε, Google και όλες αυτές τις μηχανές ε, αναφέρονται ότι ε, δεν πρέπει να είμαστε κακοί. Αυτό πρέπει να τους το θυμίσουμε. Εμείς τώρα αντιμετωπίζουμε έναν ψηφιακό καπιταλισμό και όπως κάναμε και με τον αναλογικό πρέπει να προχωρήσουμε και να ε, ελέγξουμε και τον ψηφιακό καπιταλισμό και να αντιμετωπίσουμε ε, όλα, ε, όλες αυτές τις απειλές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, απέναντι ε, σε αυταρχικούς ηγέτες. Οι, οι συνέπειες για μένα είναι σαφείς. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, γιατί είναι ένα καυτό θέμα, αν πρέπει να έχουμε μια δημόσια ευρωπαϊκή ε, πλατφόρμα η οποία θα αριθμίζεται με τρόπο ευφυή, ε, δεν θα είναι όπως τα δημόσια ε, μέσα και τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, αλλά θα ε, αναφέρεται σε συστήματα όπως τα αμερικανικά μονοπόλια. Ακόμα και η New York New York Times ε, δεν εξαιρούνται ε, από τα προβλήματα και πάρα πολλοί ε, Αμερικανοί επισημαίνουν κινδύνους στη δημοκρατία. Το Google και το Facebook είναι de facto νέου τύπου μιμιέ και πρέπει να ρυθμίζονται, χρειάζονται ίσοι κανόνες του ανταγωνισμού μεταξύ παλιών και καινούριων ε, ε, ε, έχουμε και την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο όπου θα πρέπει να δούμε τον ενεργητικό και τον παθητικό του ρόλο και σε πολιτικό επίπεδο να το ρυθμίσουμε. Η Μαρκρέτε Βεστάγκερ, η Επίτροπος Ανταγωνισμού, το Google, το Facebook ε, και άλλους τους ε, ε, αναγκάζει να πληρώσουν φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και την εμπορική χρήση των άρθρων στον τύπο και όλο αυτό το, το πρόβλημα των copyrights πώς έχει το copyright όταν αυτά ανεβαίνουν σε πλατφόρμες δεν μπορούμε να κινούμεθα σε ιδιωτικό επίπεδο θα πρέπει να πληρώνουν φόρους και θα πρέπει να πληρώνουν για άδειες. Επίσης, δεν χρειάζεται γενικό φίλτρο, ε, δεν είναι θέμα αυτό ε, ε, πρόβλημα και ε, δεν είναι το θέμα ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία του τύπου. Ε, το σημαντικό είναι ότι χρειάζεται παντού διαφάνεια. Υπάρχουν κάποια πιλωτικά προγράμματα που θα το ρυθμίσουν αυτό. Χρειάζεται πολιτική δράση. Γιατί είμαστε οι υπερήφανοι Ευρωπαίοι νομοθέτες και πρέπει να αναλάβουμε το έργο μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και σίγουρα ε, θα μας ε, φανούν πάρα πολύ χρήσιμα τα όσα ακούσαμε γιατί ε, η πολιτική έχει μείνει ανενεργή όσον αφορά τα θέματα αυτά. Το ζήτημα των κοινωνικών δικτύων αυτών, το φαινόμενο των fake news, των ψευδών ειδήσεων, έχει μολύνει ε, όλη την ε, παραδοσιακή ε, πληροφόρηση. <laughs> Δηλαδή σήμερα πλέον ακόμα και στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο γραπτό τύπο υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Στην ουσία δηλαδή λίγο έχουν συνηθίσει όλοι να μην εξακριβώνουν, να μην τσεκάρουν και διασταυρώνουν τις πηγές τους. Αυτό το οποίο συμβαίνει ακόμα ε, ε, στα παραδοσιακά ε, μέσα ενημέρωσης είναι ενδεχομένως κάποια παρεμβολή που δεν γίνεται τόσο στα ψηφιακά δίκτυα και αφορά το κοινό. Το κοινό έχει συνηθίσει να βλέπει με διαφορετικό τρόπο τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης όσον αφορά ας πούμε το ποιοτικό επίπεδο. Ξέρουμε στις γερμανικές τις ε, ε, στις ε, ε, γερμανικές ας πούμε εφημερίδες το κοινό ξέρει ποια είναι η εφημερίδα η οποία είναι πιο αξιόπιστη κτλ. Αλλά στα δίκτυα το, ο αριθμός των κλικ είναι, αυτά, είναι αυτός ο οποίος μετράει, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο σημαντικός. Εκεί θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μας βοηθήσετε, θα πρέπει να μας δώσετε κάποιες ιδέες έτσι ώστε να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο να προχωρήσουμε σε αλφαβητισμό όσον όσον αφορά τα νέα μέσα, ε, να μάθει ο κόσμος να εκπαιδευτεί. Εάν δεν παρέμβουμε ε, στην αρχή της ε, πρόθεσης του fake news, ε, μετά είναι πάρα πολύ αργά. Δεν έχει καμία έννοια να παρέμβουμε αργότερα, όταν έχει ήδη αρχίσει να κυκλοφορεί. Υπάρχει βεβαίως η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία πριν από 16 χρόνια και τότε το ηλεκτρονικό εμπόριο ήταν ακόμα στα σπάργανα, για να μην πω ήταν ακόμα στο μεσαίωνα. Ε, η Σίλβια Κώστα αναφέρθηκε προηγουμένως ε, ε, στο πρόβλημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, τον, έλεγχο δηλαδή των πλατφορμών. Μας λένε ότι αυτό είναι ένα είδος λογοκρισίας, αλλά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος βάζει τις ειδήσει. Δεν είναι άγρια δύση εδώ, δεν είναι στην πλατφόρμα, δεν είναι άγρια δύση, δεν είναι Far West. Ευχαριστώ. Προχωρούμε στα άλλα μέλη, μέγιστος χρόνος 2 λεπτά. Η κυρία Χιμένες. Ζητώ συγγνώμη, έφτασα λίγο αργά, δεν άκουσα από την αρχή, αλλά άκουσα τον κύριο Μαρκιόρη. Ε, αναφερθήκατε σε blue lights. Όχι, ο κύριος blue lies. Α, ναι, blue lies, ναι. ψέματα. Μπλε ψέματα. Ε, τα οποία δικαιολογούνται ε, επειδή τα προωθεί μια ομάδα. Τι να σας πω, στην Καταλωνία, γιατί εγώ θα μιλήσω για αυτά που ξέρω και τα δικά μου, έγινε μια εκστρατεία όπου υπόθηκαν πράγματα ψευδή ε, ο, μετά έγινε γνωστό πλέον και απεδείχθη ότι ήταν ε, ε, ψευδείς οι ειδήσει, αλλά ο κόσμος διαμόρφωσε γνώμη και πήρε απόφαση βάσει αυτών των ε, ψεμάτων και θα ήθελα λίγο να μου το εξηγήσετε αυτό έτσι ώστε να καταλάβω κι εγώ ακριβώς πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα στη δικιά μου περιοχή. Ο συνάδελφος Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω, ποιοι είναι οι θεματοφύλακες της αλήθειας. Το ρωτώ αυτό γιατί το φαινόμενο των fake news δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα αυτούσιο ανεξάρτητο φαινόμενο, αλλά λειτουργεί μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Όταν μιλάμε για αρχές, ρυθμιστικές αρχές, τι εννοούμε. Ένας, ο Πίρτς Όμπσπορν, ένας ε, ε Άγγλος ε, συγγραφέας, ε, έγραψε ένα βιβλίο για το πώς σκέφτεται ο Τραμπ. και έχει γράψει και άλλες, εκθέσεις, και άλλες αναφορές με αυτό το θέμα. Γιατί τον αναφέρω. Γιατί στις προεκλογικές εκστρατείες το σύστημα των αλγορίθμων που ανέφερε ο κύριος Χένριξ χρησιμοποιούνται και για αυτό το σκοπό. Ε, ζητάμε αλλαγές ε, στη, στα κρατικά μημία που πρέπει να προστατευόνται και να παρέχουν σωστή ενημέρωση στην κοινή γνώμη. Τι διασφαλίσεις ε, πρέπει να έχουμε για να γίνει αυτό, πώς μπορούμε να το κάνουμε. Επίσης, Πώς μπορούμε να συσχετίσουμε αυτό που γίνεται με τα fake news και τη χειραγώγηση σε διεθνές επίπεδο. Για παράδειγμα, τις ε, κατηγορίες ότι η Ρωσία παρεμβαίνει στην εκστρατεία για τον Brexit ή στην προεκλογική εκστρατεία στις Ηνωμένε Πολιτείες ή σε άλλες προεκλογικές εκστρατείες. Ε, έχουμε τέτοια fake προφίλ. Ε, ερωτώ λοιπόν ποιον θα εμπιστευτούμε να τον κάνουμε θεματοφύλακα και ρυθμιστική αρχή για να φροντίσει να υπάρχει αλήθεια για όλους. Ευχαριστώ. Η κυρία Σιόιντροβα. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Συνεχίζω μετά τις ερωτήσεις σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσω με τη λεγόμενη λογοκρισία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην οδηγία για την αναθεώρηση για των οπτικοακουστικών ζητεί κάποια περιεχόμενα να απαλληφθούν. Ε, ε, ε, δηλαδή ρητορική μίσους, παρακίνηση σε ριζοσπαστικοποίηση, τρομοκρατία. Αυτά τα περιεχόμενα πρέπει να απαλληφθούν. Αλήθεια είναι ότι πολλοί λέ, μας επικρίνουν και λένε εδώ έχουμε λογοκρισία κλπ. Θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε οποιοδήποτε δημοσιεύει, οποιασδήποτε ειδήσει θα πρέπει να είναι επαληθεύσιμο μη πηγή. Μπορεί να είναι δυσάρεστες ειδήσει για κάποιους προσωπικά για μένα, αλλά αν δεν υπάρχει ε, η πηγή, ποιος θα είναι υπεύθυνο. Αυτή είναι ο κίνδυνος της δημοκρατίας. Υπάρχει η ελευθερία, αλλά δεν υπάρχει ευθύνη. Ας υπάρχει λοιπόν ε, ελευθερία, αλλά ο καθένας να αναλαμβάνει την ευθύνη των γραφωμένων του. Και το λογικό ερώτημα που προκαλείται είναι το ανώνυμο περιεχόμενο μήπως δεν πρέπει να δημοσιεύεται, διότι αν δημοσιεύεται δεν μπορούμε πια να επαληθεύσουμε, να εντοπίσουμε ποιος είναι αυτός που στέλνει τα συγκεκριμένα μηνύματα. Ο καθένας μπορεί ατιμωρητή δηλαδή να δημοσιεύει ό,τι θέλει. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γραμματικάκης. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή συζήτηση Χαίρομαι κύριε Πρόεδρε γιατί πράγματι εξελίσσεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ή σχόλιο. Ε, το πρώτο σχόλιο. Ξεχνάμε ότι δεν είναι καινούριο πράγμα τα fake news. Είναι πολύ παλιό, όσο ίσως η ηλικία της ανθρωπότητας. Το καινούριο φαινόμενο είναι ότι έχουν πυκνώσει είναι δύσκολο να διευκρινιστεί η αλήθεια τους. Επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. Να θυμίσω όμως ότι πριν από 30-40 χρόνια ο Wells στην Αμερική έκανε μια εκπομπή όπου περιγραφόταν η εισβολή εξωγήινων στη Νέα Υόρκη. Και αυτό προκάλεσε βέβαια τον τρόμο μέχρι ότου ο Wells διευκρίνησε ότι ήταν ένα αστείο. Είναι fake news αυτό ή όχι αλίμονο αν χάσουμε και την ψυχαγωγία τέτοιου είδους. Η δεύτερη παρατήρηση άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την κατάταξη που κάνατε και τους ορισμούς που δώσατε στα fake news. Ε, εγώ θα βλέπα ένα άλλο τρόπο να τα κατατάξει κανένας. Αν είναι εύκολα επιβεβαιώσιμα ή όχι. Φερρυπίν αν διαβάσαμε στο Google ότι ένα μήλο αρχίζει να πηγαίνει όχι προς τη γη αλλά προς το διάστημα μόνο του εντάξει αυτό το ξέρουμε το διαψεύδουμε αμέσω. μια άλλη όμως είδηση που μιλάει για χιλιάδες θύματα στη Νότιο Αμερική για παράδειγμα πρέπει να έχουμε πολλές πηγές πληροφοριών για να δούμε αν είναι αλήθεια ή όχι την έκταση του ψέματος. Και υπάρχουν βέβαια και ειδήσει που είναι μάλιστα πολύ της μόδας για παράδειγμα οι φημολογούμενες ή αληθινές σεξουαλικές παρενοχλήσεις που είναι αδύνατον προφανώς να βρει κανένα στην αλήθεια. Μια κατάταξη λοιπόν παρομοίου είδους πόσο εύκολα επιβεβαιώσιμη ή όχι είναι μια ψευδής είδηση θα μας φώτιζε πάρα πολύ αυτό που ψάχνουμε. Γιατί νομίζω ότι είμαστε στη φάση που περιγράφουμε πολύ καλά το φαινόμενο έστω πολλές φορές με διανοητική υπερβολή, αλλά οι λύσεις δεν φαίνονται ακόμα ορατές. Ε, μια σαφής απάντηση, αλλά η καλύτερη παιδεία μπορεί να το λέμε εμείς εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού, αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολο να γίνει και ισχύει σαν ένα fake news, το καλύτερη παιδεία. Δεν γίνεται. Vielen σας ευχαριστώ πολύ και καθηγητά και πριν λησμονήσω να απευθύνω το καλό ορίσατε στην ομάδα επισκεπτών. 20 ασκούμενοι και ασκούμενες της Γενικής Διεύθυνσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις μεταφράσεις. Νέοι και νέες μεταφράστριες δηλαδή. Και ελπίζω ότι σας προσφέρει και κάποια γνώση η παρακολούθηση της ε, συνεδριάσεώς μας. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Σαβίνη, δύο λεπτά και μετά θα λάβουν το λόγο πάλι οι εμπειρογνώμονές μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μας δίνετε το λόγο στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Πράγματι, οι ιδέες που προέκυψαν από τις παρεμβάσεις και τους, ε, των ομιλητών και των ε, βουλευτών έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και η Κομισιόν με ενδιαφέρον τα σημειώνει όλα αυτά. Ιδιαίτερα τώρα που ο Επίτροπος Γκαμπριέλ η Επίτροπος ανακοίνωσε πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των fake news την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ξεκινήσει δηλαδή μια δημόσια διαβούλευση η οποία θα συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου που είναι ήδη ανοιχτή τώρα και όλοι μπορούν να καταθέσουν απόψεις και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το Φεβρουάριο και μετά θα δημιουργηθεί μια ομάδα υψηλού επίπεδου η οποία με τρόπο αναλογικό θα αντικατοπτρίζει τις διάφορες συνιστώσεις που συνθέτουν το πρόβλημα και τη λύση του ίσως. Μια ομάδα υψηλού επίπεδου που θα παρουσιάσει με τρόπο ισορροπημένο το έργο των πλατφορμών, της έρευνας, του δημοσιογραφικού κόσμου και των ε, οργανώσεων της, ε, των πολιτών. Τώρα λοιπόν ακούμε και θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα πώς το φαινόμενο αυτό διαμορφώνει με τρόπο αρνητικό την κοινή γνώμη και να δούμε βέβαια και τη ζημία που προκαλεί αυτό το φαινόμενο. Αυτό είναι στο προσκήνιο όλων των συζητήσεων και αυτό φάνηκε και σήμερα. Ε, αναδεικνύεται η ανάγκη άμεσης δράσης και ορισμένες ιδέες και στόχοι είναι ξεκάθαροι στην Κομισιόν όπως ε, η διαφάνεια, η ορατότητα, θέματα που αφορούν τους αλγορίθμους ε, και το πώς ε, προβάλλονται περιεχόμενα σε περιβάλλον online όπως και διαφάνεια όταν πρόκειται για τις χρηματικές ροές που πολλές φορές στηρίζουν τη διάδοση παραπληροφόρησης ε, ε, με κακόβουλο τρόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και ελπίζω ότι η παρούσα συνάντηση μπορεί να επιτρέψει την απόκτηση γνώσεων και του από πλευρά Κοινοβουλίου αλλά και από πλευρά από πλευράς συγγνώμη, Επιτροπής. Ας δώσω πάλι το μικρόφωνο στους εμπειρογνώμονες μας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε όλοι σε όλες τις ερωτήσεις. Επιλέξτε κάποια ερώτηση που θα θέλατε να απαντήσετε. Και το λόγο μπορείτε να λάβετε ε, ας πούμε για δύο-τρία λεπτά ο καθένας. Παρακαλώ λοιπόν να περιοριστείτε στα ουσιώδη όπου θεωρείτε ότι πραγματικά πρέπει να απαντήσετε. Ο κύριος Μαρκιόρη. Είναι κρίμα, κρίμα. Τόσο πολλές ερωτήσεις, τόσο λίγος χρόνος. Όλες ε, είναι πολύ σημαντικές οι σκέψεις που εκφράσατε. Μπορεί να συνοψίσει κανείς με λίγα λόγια, ωστόσο. από νεαρά παιδιά τα άκουσα αυτό, αυτά, που τα νεαρά, τα πολύ μικρά παιδιά είναι και το πιο δύσκολο ακροατήριο, γιατί αμέσω ρωτούν γιατί. Και αμέσω πια, ακόμα πιο σημαντικό, γιατί όχι, το οποίο τρομοκρατεί τον ε, εμπειρογνώμονα, διότι ό,τι τους πείτε δεν το θεωρούν ε, αυτονόητο και διαστρωματωμένο κλπ. Εμείς ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι διαστρωματωμένη. Σημαίνει ότι έχουμε κάποια ιεραρχία και υπάρχει και μια αδράνεια απέναντι στι αλλαγέ. Τι σημαίνει αυτό τώρα πιο συγκεκριμένα. Α πάρουμε τους αλγορίθμους. Η διασπορά των ε, ψευδών ειδήσεων που γίνονται viral φαίνεται σαν να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτε, διότι αυτό είναι το διαδίκτυο. Έτσι λειτουργεί το διαδίκτυο, λέει, σα λένε πολλοί. Όχι, όχι, δεν είναι αναγκαίο να λειτουργεί έτσι το διαδίκτυο με αυτόν τον τρόπο. Εμεί το κάνουμε να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε όμω και να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργία. Απλό είναι. να παρεμποδιστεί αυτή η viral διασπορά των ειδήσεων. Όχι όμως να λογοκρίνεται, γιατί εάν λογοκρίνεται κάτι, μπαίνετε σε κάπως ε, δύσκολα νερά. Λογοκρισία σημαίνει όχι, σε βγάζω, δεν έχεις το δικαίωμα να πεις τίποτα. Όμως άλλο πράγμα είναι ο πολλαπλασιασμός που μπορεί να μην εμπιστεύομαι. Δεν έχει σχέση με τη λογοκρισία. Ο, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το διαδίκτυο είναι ότι ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει και αυτό να πολλαπλασιάζεται επάπειρον. Αυτό όμως δεν είναι ελευθερία, είναι ανοησία. Διότι το διαδίκτυο δεν γεννήθηκε για να διευκολύνει τέτοιου είδους καταστάσεις. Το διαδίκτυο αρχικά μπορεί να πει κανείς γιατί έχουμε όλους αυτούς τους hacker τα προβλήματα ε, των ε, της ασφάλειας. Αρχικά το διαδίκτυο δημιουργήθηκε για στρατιωτική χρήση και ήταν απόλυτα ασφαλέ. Μετά άνοιξε βέβαια στο κοινό. Και τώρα τι κάνουμε, αλλάζουμε το διαδίκτυο. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πρωτοκολλά ώστε να γίνει πιο ασφαλέ. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει για την ελευθερία πληροφόρηση. Το δίκτυο άρχισε με ένα συγκεκριμένο τρόπο με πολύ λίγου που διοχέτευαν πληροφορίε και δεν υπήρχε θέμα fake news δεν υπήρχαν καν news αρχικά στο διαδίκτυο. Τώρα όμως έχουμε φτάσει να έχουμε τα προβλήματα αυτά. Υπάρχει λύση. Γιατί όχι. Αλλάζουμε το μοντέλο χωρίς να λογοκρίνουμε αλλά προλαμβάνουμε ε, τον, τον άπειρο πολλαπλασιασμό. Δύο λεπτά για να απαντήσω σε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Θα είναι πρόκληση. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε τρεις ερωτήσεις. Αν κάτι σας φαίνεται σαν τύπος, σας μυρίζει σαν τύπος, τότε μάλλον είναι τύπος. Έχουν τα δικά τους πρότυπα ελευθερία λόγου και στα κοινωνικά μέσα. Ισχύει. Έχουν στην πραγματικότητα εφημερίδες μαζικής κυκλοφορίας και ε, δικτυακές πύλες ελευθερία λόγου. Αυτό σημαίνει. αρχίζει το blog όπου θέλει καθένας και μπορεί να λέει ό,τι θέλει με αυθαίρετο τρόπο. Τα κάνουν αυτά ήδη. Αν ήμουν εγώ λοιπόν Ευρωπαϊκή Ένωση θα πήγαινα στον ΩΣΑ, στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλους μεγάλους σοβαρού φορεί να πω ότι κοιτάξτε αποτελεί παγκόσμια πρόκληση πλέον η ελευθερία στο διαδίκτυο και αν ήμουν εγώ θα έλεγα είστε τώρα στην πραγματικότητα συντάκτες μαζικών πρακτορείων παροχής πληροφοριών. Δικό σας είναι το πρόβλημα αν έχετε δύο εκατομμύρια δημοσιογράφους. Έχετε εσείς εδώ την εξουσία, εσείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είσαστε τίποτα, κανένα αυθαίρετος φορέας. Ανάμεσα σε ένα πολιτικό θεσμό και οποιοδήποτε άλλο φορέα, εσείς ισχύετε. Έχετε την, την ισχύ και τίποτα δεν μπορεί να σας απαντήσει. Ακόμα και αν είστε liberal με την έννοια του απόλυτα φιλελεύθερου μπορεί να πρέπει να ρυθμίσετε γιατί τελικώ η αγορά δεν τα ρυθμίζει από μόνη της. Και αν δεν ρυθμίσετε νομοθετικά εσείς θα καταλήξετε να έχετε από τη μια του τεσπεράντος που κάνουν ό,τι θέλουν και τον ελεύθερο τύπο από την άλλη μεριά που δεν έχει την ελευθερία ωστόσο να πει ακριβώς ό,τι θέλει διότι είναι υποχρεωμένος να τηρεί πρακτικές, βέλτιστες πρακτικές της δημοσιογραφίας, πρότυπα κλπ. Και αν ήμουν εγώ ε, στη θέση σας και μου λέγατε ότι χρειάζεται checks and balances για επαλήθευση πληροφοριών. Διαβάστε τον κώδικα διοντολογία της Αμερικανικής Ένωσης Δημοσιογράφων που λέει «Ακολουθήστε την αλήθεια όσο μπορείτε, κρίνετε τις πηγές σας και συνεχίστε στην βάση αυτή». Έχουν ένα κώδικα για την αλήθεια στη δημοσιογραφία. Αυτά να χρησιμοποιήσετε. Και στα υπόλοιπα βάλτε να λειτουργήσουν οι επιστήμονες. Για ό,τι αφορά τα κιανά ψέματα, τα blue lies, η κοινωνική ψυχολογία, ε, βέβαια την έχουμε από πάντα, τώρα έχει επιταχύνει η κοινωνική ψυχολογία και κυριολεκτικά και με κάποια έμφαση. Αλλά έχω να πω το εξή. Αυτά τα φαινόμενα, τα μπλε ψέματα και όλα τα σχετικά, σας οδηγούν να αλλάξετε πεπιθήσεις και να αλλάξετε συμπεριφορά που στην ουσία βασίζονται σε ένα είδο δυναμική ομάδα. Αν ήμουν Ευρωπαϊκή Ένωση θα διέθετα χρήματα να κάνω μελέτε για την κοινωνική ψυχολογία στο διαδίκτυο. Ίσως προ τα εκεί. Να μα δώσετε κάποια λεφτά και προ εμά εδώ τους επιρογνώμονες του πάνελ. Και τα fake news υπάρχουν από τότε που υπάρχει ανθρωπότητα, δεν είναι τίποτα το νέο. Αυτό που είναι νέο είναι ότι έχουμε τώρα μια διάδοση που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Από την άποψη αυτή είναι απολύτως νέα τα πράγματα αυτά για όλους. Αλλά να τονίσω ένα επιχείρημα. Ολόκληρη αυτή η ιδέα ότι η πλατφόρμα στο Facebook και Google κτλ. είναι απολύτως ελεύθερη. Όχι, δεν είναι. Δεν μπορείς να πεις ότι θέλει. Όχι, καθόλου. Γιατί δεν χρησιμοποιείτε ακριβώ αυτό το επιχείρημα και να πείτε τώρα που εσείς είστε απευθυνόμενοι στους άλλους δηλαδή εκδότε τεράστιων ειδήσεων, να κινηθείτε. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος πολύ σημαντικός. Χωρίς μικρόφωνο δεν ακούν οι διερμηνείς. Με μικρόφωνο παρακαλούμε. Εγώ θα ήθελα να χωρίσω το ε, ε, θέμα σε δύο τμήματα. Το πρώτο αφορά την πληροφόρηση και το άλλο αφορά την γεωπολιτική η διάδοση των ε, πληροφοριών αφορά το πρώτο τμήμα με την έννοια που το έθεσαν οι συνάδελφοι και νομίζω ότι αυτό μπορεί να λυθεί με τον ένα τον άλλο τρόπο. Εγώ προβληματίζομαι ιδιαίτερα με το δεύτερο σκέλος γιατί τα ψεύτικα νέα ε, στο ε, διαδίκτυο όταν έχουν σκοπιμότητες πολιτικές, όταν κάποιοι υποστηρίζουν και προωθούν τα fake news, δημιουργούν τα sites, ε, τα σημεία στο ίντερνετ, τους ανθρώπους ε, που ε, θα προωθήσουν τα νέα αυτά. Στην Βουλγαρία βλέπουμε κάθε μέρα καινούρια μέσα, μέσω των οποίων διαδίδονται αυτές οι ειδήσει. Το πρόβλημα λοιπόν, το δεύτερο σκέλος δηλαδή, του προβλήματος του γεωπολιτικό είναι λίγο πιο ευαίσθητο και δεν είμαι και τόσο αισιόδοξο. Υπάρχουν πολιτικά ζητήματα, ε, ε, θέματα ταυτότητας, ε, θέματα επιλογών, θρησκευτικών κτλ. Και όταν κανείς θέλει να μοιραστεί κάποιες ιδέες με ανθρώπους που έχουν τα ίδια πιστεύω, που έχουν την ίδια θρησκεία, εκεί ο έλεγχος είναι πολύ πιο δύσκολος και νομίζω ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο ε, ε, ε, αναφερόμαστε στην πολιτική, ακόμα και στα πανεπιστήμια. Από τη μία μεριά λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ανάγκες, οι ανάγκες του κόσμου, οι δημόσιες ανάγκες ε, για τη διαμόρφωση του πολιτικού λόγου και από την άλλη ε, πώς μπορούν να επηρεαστούν οι ανάγκες. Εγώ τώρα βλέπω ε, κάποιες ενδιαφέρουσες κινήσεις που αφορούν κατά κάποιο τρόπο την άτυπη πολιτική. Εάν δει κανεί τα συγγράμματα της συγκριτικής ε, ε, πολιτικής, ε, τότε βλέπετε, θα δείτε ότι υπάρχει εστίαση σε, πιο, σε κάποια βασικά στοιχεία ε, και ε, ε, γίνεται αναφορά στα σωστά στοιχεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί η πολιτική. Ακριβώς το αντίθετο κάνουν τα fake news. Τώρα βλέπουμε και παραδείγματα αριστείας στην δημοσιογραφία και ίσως αυτό πιο πολύ να το βλέπουμε στην Ευρώπη αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι προφανές και εύκολο να το βρει κανείς σε άλλα σημεία. Το σημαντικό επομένως δεν είναι νομίζω ε, να ε, μάθεις τους ανθρώπους ε, να βλέπουν ποιος είναι ο άριστος και σωστός δημοσιογράφος αλλά να του δώσεις τη δυνατότητα να μάθει να διαβάζει με κριτικό τρόπο τις ειδήσει. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την πρώτη πολύ διαφωτιστική συζήτηση. Ε, είχαμε μια πολύ ζωντανή συζήτηση και πάμε τώρα στο δεύτερο γύρο, στο δεύτερο πάνελ. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε εδώ τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, καθηγητή στο MIT, τη Βοστόνη, ο οποίος ε, θα μας μιλήσει για τις ε, επιστημονικές και τεχνολογικές προσεγγίσεις που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν για να προσεγγίσω με τα fake news και καλωσορίζω και τη μοναδική κυρία ανάμεσά μας, την κυρία Καρολίν Σουάρτσε που είναι συνεργάτρια σε ένα ερευνητικό κέντρο μη κερδοσκοπικό στο Βερολίνο που λέγεται Corrective και ασχολείται με την αποκάλυψη των fake news και θα μας ε, μιλήσει και για πρακτικά θέματα πόσο συχνά ανακαλύπτονται τα fake news, πώς θα αντιμετωπίζουμε και πώς θα ε, προβάλλουμε. Να δώσω πρώτα το λόγο στον καθηγητή κύριο ε, Δασκαλάκη για 10 λεπτά και μετά στην κυρία Σουάρτς. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Μπορώ να έχω το κλίκαρα. χειριστήριο. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, κυρίως γιατί δεν υπάρχει σαφής ορισμός του τι είναι fake news. Είναι δύσκολο να προτείνουμε ορισμό χωρίς να μπούμε σε φιλοσοφικά θέματα του τι είναι γεγονός, τι είναι αλήθεια κλπ. Σίγουρα ένας ορισμός εργασίας είναι ότι τα fake news είναι η σκόπιμη ε, λάθος αναπαράσταση ενός συμβάντος, ε, λάθος παρουσίασή του, όπως φαίνεται εδώ αριστερά, ή μια πληροφορία εντελώς κατασκευασμένη με στόχο την εξαπάτηση του κόσμου. Όπως ακούσαμε ήδη, είχαμε και στο παρελθόν fake news, δεν καινούριο φαινόμενο αυτό. Οπότε αυτό που είναι το κρίσιμο θέμα προς συζήτηση σήμερα είναι η άλλη συνιστόσα του fake news, δηλαδή ο τρόπος διάδοσης. Ο ορισμός του fake news θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τον τρόπο διάδοσης. Και τα fake news θα πρέπει να, να, να, να, να ε, επεκταθούν για να συμπεριλάβουν και την ενορχιστρωμένη προώθηση ε, πραγμάτων ε, με τρόπο που φαίνεται ότι η πρόθεση αυτή γίνεται από πραγματικούς ανθρώπους. Αν φαίνεται ότι είναι από πραγματικούς αλλά είναι κατασκευασμένο, αυτό συνιστά fake news. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το πώς εξαπλώνονται τα ε, fake news και να δούμε και κάποιες τεχνικές προσεγγίσεις για να καταπολεμήσουμε ίσως τα fake news. Τα κοινωνικά bots και οι ψεύτικοι λογαριασμοί στο δίκτυο παίζουν τεράστιο ρόλο στη διάδοση των fake news οργανωμένες εκστρατείες, ε, χρησιμοποιούν ομάδες κοινωνικών bots ε, και ψεύτικους λογαριασμούς για like, για share, για retweet. Ε, υπάρχει εδώ μια click farm, μια ομάδα δηλαδή που κλικάρουν και φαίνεται σαν να είναι ένας πραγματικός άνθρωπος που αλληλεπιδρά. Ο στόχος λοιπόν της χρήσης bots και click farms εδώ ε, είναι να ε, προκαλέσουμε ε, αλγορίθμους σε όλα αυτά τα facebook κλπ που θα καθορίσουν ποιες πληροφορίες παίρνουν την προτεραιότητα και ποιες ειδήσει είναι ελκυστικές και αξίζουν να προωθηθούν ενώ είναι fake news. Μπορεί να, είναι, να μην είναι στον πυρήνα των κοινωνικών δικτύων, μπορεί να είναι σε περιθωριοποιημένα, αλλά εξαπλώνονται και εν μέρη συνδέονται και με νόμιμους και πραγματικούς χρήστες. Και γι' αυτό είναι δύσκολο ε, να ε, είναι πάντα πραγματικοί άνθρωποι. Επίσης, είναι, τα fake news είναι συνδεδεμένα με τους χρήστες και μπορεί κανείς και να αγοράσει ε, από τους λογαριασμούς αυτούς ε, περιεχόμενα. Επίσης, ε, μπορεί κανείς, αν πληρώσει, να προσελκύσει και κάποια διασημότητα να ασχοληθεί μαζί σας. Και αυτό είναι δύσκολο. Αν δηλαδή πληρώνετε ένα πραγματικό άτομο να ε, συμμετέχει στο λογαριασμό σας, ε, αυτό είναι δύσκολο να αποδειχθεί ως ε, ψευδές περιεχόμενο. Εδώ κάνω μια προσπάθεια να συνοψίσω την εξάπλωση των fake news. τα fake news μπαίνουν μέσα από κάποια γωνία στο κοινωνικό δίκτυο και με προκλητικό περιεχόμενο προκαλεί εντατικό clicking, sharing, retweeting και κοινωνική ε, ενασχόληση. Βλέπουμε την είσοδο, αρχίζουν τα κλικ ε, και μετά ε, αυτή η συμμετοχή ενισχύει ε, αυτό που θεωρείται ως καλό περιεχόμενο και σε άλλα κοινωνικά μέσα. Και ε, έτσι έχουμε ακόμη μεγαλύτερη θέαση και έτσι πολλαπλασιάζεται ε, η εμβέλεια των fake news. Και βέβαια τα διαφημιστικά έσοδα είναι μεγάλα, αυτός είναι ένας λόγος που έχουμε fake news και επηρεάζουν με το περιεχόμενό τους πολιτικές ιδεολογίες ε, μπορεί να δημιουργήσουν ε, ε, διαμαρτυρίες, να προκαλέσουν εκλογές ακόμα. Αυτό μπορεί να συμβεί. Πώς μπορούμε να ανοιχνεύσουμε τα fake news. Η ανοιχνεύση τους είναι πάρα πολύ δύσκολο καθήκον ακόμα και για εκπαιδευμένους ελεγκτές αληθινών δεδομένων. Δυστυχώς τώρα τεχνικά δεν ε, είναι δυνατόν αυτόματα να εντοπίζουμε τα fake news με κάποια ε, ακρίβεια, ας πούμε 90%. Οπότε αυτό είναι ένα σύνθετο καθήκον το οποίο αφορά την πηγή των ε, ειδήσεων και έχει να κάνει και με την προηγούμενη λειτουργία των πηγών ειδήσεων ε, έχει να κάνει με την ε, παρουσία τίτλων ελκυστικών, την ποιότητα της γλώσσας, ε, το περιεχόμενο άλλων άρθρων του ιδίου θέματος που έχουν δημοσιευτεί από αξιόπιστες πηγές. Εκεί υπάρχει μια σύγχυση. Υπάρχουν ε, θέματα όπως οι αλγόριθμοι, η τεχνητή νοημοσύνη, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, ε, ε, γλωσσολογία, επιστήμη δικτύων, ψυχολογίας που όλα αυτά ενέχονται. Δεν είναι με την τωρινή τεχνολογία να τα με τα fake news. Υπάρχουν όμως τρόποι να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να βοηθήσουμε τον προσδιορισμό ενός fake news. Ε, υπάρχουν τεχνολογίες για να συγκρίνουμε το σώμα ενός άρθρου με τον τίτλο του, ε, να καθορίσουμε την ποιότητα της σύνταξης και της γραμματικής ένα άρθρο, ε, να εντοπίσουμε εμπριστική γλώσσα, να κάνουμε ανάλυση συναισθημάτων. Υπάρχουν δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης προσεγγίσεις που θα μας βοηθήσουν αυτά χρησιμοποιούν αυτοί που επαληθεύουν τα ε, γεγονότα. Υπάρχει επίσης τεχνολογία και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί αυτό που κάνει μια είδηση fake δεν είναι μόνο το περιεχόμενο, αλλά και διαδικασία εξάπλωσης που είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχουν λοιπόν αλγοριθμικές προσεγγίσεις που ε, δείχνουν το ρόλο των ε, κοινωνικών bot. Βλέπετε εδώ πώς γίνεται είσοδος από τη γωνία ενό κοινωνικού δικτύου. Υπάρχουν λοιπόν αλγόριθμοι δικτύων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να δούμε αν υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι τρόποι ε, χρησιμοποίησης και ε, προβολής fake news. Λοιπόν, είπαμε για την ανείχνευση με την τωρινή τεχνολογία. Είναι σημαντικό όμως να πιάσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του, να αλλάξουμε δηλαδή την τεχνολογία, ούτως ώστε η εξάπλωση των fake news να δυσχεραίνεται, να, να δυσκολέψει. Ήδη υπάρχουν κάποια μέτρα που ε, αναστέλουν την ε, διάδοσή τους και την κερδοφορία των πηγών, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με το χρήμα. ο Google έχει κάνει ε, blacklist καταχρηστικών websites και τώρα εφαρμόζει αλλαγές στην μηχανή αναζήτησης για να μην μπορέσει να φάσει ψηλά το περιεχόμενο που δεν είναι αξιόπιστο. Οι Facebook και Twitter έχουν μηχανισμούς για την αναφορά, εντοπισμό και αναστολή των καταχρηστικών λογαριασμών. Οπότε ένα πολύ ισχυρό μέσον είναι να χρησιμοποιήσουμε τους χρήστες για να ε, επισημάνουν κάποιο fake news, δηλαδή μπορεί να ε, σηκώσει μια κόκκινη σημαία ας πούμε. Βέβαια αυτό έχει και αυτό τις δυσκολίες του, γιατί αν δεν γίνει με τρόπο ευφυή και με σίγουρο τρόπο Ούτως ώστε, πρέπει να γίνει με τρόπο ε, ε, τέτοιο ώστε να μην σηκώνουν κόκκινο σημαίακι οι χρήστες όταν βλέπουν κάτι με το οποίο διαφωνούν. Η Wikipedia μπορεί να βοηθήσει για το πώς μπορεί να εφαρμοστούν όλα αυτά. Επίσης, ε, θα ήταν εάν ε, ε, υπάρξει προειδοποιητικό μήνυμα σαν κόκκινη σημαία όταν ένα άρθρο θεωρηθεί αμφιλεγόμενο θα μπορούσε να είναι ένα μέσον. Η αξιοπιστία ενός άρθρου σχετίζεται επίσης με την αξιοπιστία της πηγής και υπάρχουν μηχανισμοί διαφοροποίησης μεταξύ αξιόπιστων και μη αξιόπιστων πηγών ειδήσεων. Βέβαια δεν υπάρχει καθολική συμφωνία σχετικά με το ποιες ε, πηγές ειδήσεων είναι αξιόπιστες, επειδή πολλές φορές ε, παίζουν ρόλο οι πολιτικές συμπάθειε, ποιο θα είναι αυτός που θα κρίνει. στι Ηνωμένε Πολιτείες οι New York Times ε, θεωρούνται αναξιόπιστη εφημερίδα από πολλούς ρεπουμπλικανούς και αντίθετα το Fox News θεωρείται πάρα πολύ αναξιόπιστο από πολλούς δημοκρατικούς αλλά αφήνοντας κατά μέρος το, τα κομματικά κριτήρια, αυτές οι πηγές είχαν συνεχή παρουσία για χρόνια και μπορεί σίγουρα να θεωρηθούν σχετικά αξιόπιστες. Από την άλλη, οι ε, πηγές των fake έχουν πολύ μικρό κύκλο ζωής, δηλαδή έρχονται και παρέρχονται. Και είναι δύσκολο γι' αυτό να ε, υπάρξει προειδοποίηση σαν red flag. Ε, μπορεί να υπάρξει επίσης και μια αξιολόγηση αξιοπιστίας. Υπάρχουν τεχνολογικές προσεγγίσεις για να μετρήσουμε την αξιοπιστία μιας πηγής. Τέλος, για να κλείσω, θα πω ότι πέρα από τεχνολογικές συζητήσεις, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, έχουμε σωστή εκπαίδευση. Ναι, με τον κόσμο ε, πέρα από τις ε, συνήθεις προκαταλήψεις η διάδοση των fake news εκμεταλλεύεται ε, μια έλλειψη διαδικτυακού γραμματισμού αν θέλετε. Οπότε μπορεί κανείς να θέλει το fake news να στηρίξει την ιδεολογία αλλά θα είναι <clears throat> λιγότερο πιθανό να το χρησιμοποιήσετε και σαν αποδεικτικό μέσο ή ας πούμε οι άνθρωποι επικρίνουν στις διαφημίσεις ε, τους ισχυρισμούς που γίνονται, δεν θα τους χρησιμοποιήσουν. Έτσι λοιπόν, ε, καλό θα ήταν να παρακολουθούμε τις τεχνολογίες και τα ε, σύνθετα οικοσυστήματα που δημιουργούν γύρω από την παραγωγή, την κατανάλωση και την κυκλοφορία της πληροφορίας. Οι <clears throat> χρήστες του διαδικτύου Καλό είναι λοιπόν να έχουν καλύτερη εκπαίδευση σχετικά με το πώ λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης και πώ οι τεχνολογίες μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο χειραγώγησης. Όλα αυτά θα μειώσουν το πρόβλημα. Ε, και σίγουρα θα πρέπει να ε, υπάρχει διαφάνεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Μάθαμε ότι τα τεχνικά μέσα φαίνεται πως μπορεί να βοηθήσουν για τον εντοπισμό των fake news, αλλά βεβαίως όχι χωρίς το ανθρώπινο χέρι. Και για το ανθρώπινο χέρι, την ανθρώπινη παρέμβαση, θα μας τα πει η κυρία Σφάρτς. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Μιλώ για την ομάδα μας, fact-checking, echt jetzt λεγόμαστε, δηλαδή πράγματι τώρα. Fact-checking, corrective που ιδρύθηκε το 2014, το Fact Checking Team υπάρχει όμως μόλις από πριν από λίγους μήνες, μέσα στο 2017. Είμαστε μια ομάδα τεσσάρων και αυτό που κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία monitoring μέσω των οποίων παρακολουθούμε τα περιεχόμενα των κοινωνικών μέσων, τα αποτιμούμε είναι και πρώην marketing tools τα οποία τα έχουμε τροποποιήσει για να χρησιμοποιηθούν για δημογραφικούς σκοπούς παρακολουθούμε και αντιδρούμε και σε ψευδείς δηλώσεις πολιτικών και άλλων φορέων παικτών που διαδίδουν τις απόψεις αυτές μέσω των ε, social media Κορεκτή φλεγόμαστε εμείς το διορθωτικό δηλαδή και είμαστε εταίρος του facebook Γερμανίας δηλαδή σε εμά φτάνουν οι ειδήσει που αφορούν το facebook για την ώρα μόνο άρθρα σε λίγο θα εξηγήσω πως γίνεται στη Γερμανία είναι δύσκολο βέβαια πρόκειται όπως είπα μόνο για άρθρα και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλα τα fact-checking teams που συνεργάζονται με το Facebook είναι ότι δεν υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή πόσες σημεούλε σηκώνονται, flagging δηλαδή, για ποια περιεχόμενα. Δεν γνωρίζουμε ποιες ιστοσελίδες ε, λαμβάνουν κάποιο χαρακτηρισμό από τους χρήστε και τα λοιπά. Έχω βάλει ένα fake slide πρώτη, πριν από τις ε, ομοσπονδιακές εκλογές για την Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή είχαμε δραστηριοποιηθεί σε συνεργασία με φοιτητές τους εκπαιδεύσαμε επί μία εβδομάδα, τους δείξαμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για fact-checking και τις διάφορες τεχνικές επαλήθευσης. Επί τρεις εβδομάδες δημοσιεύσαμε ένα newsletter που διοχετεύσαμε και σε newsrooms αλλά και σε ιδιώτες που ενδιαφέρονταν και κάθε μέρα δημοσιεύαμε τα fact checks που κάναμε, τα διαθέταμε και σε άλλους συνεργάτες, συναδέλφους, δημοσιογράφους για ενημέρωση. Δημοσιεύσαμε 77 άρθρα στην περίοδο εκείνη, 46 ήταν κλασικά fact checks, όπου δηλαδή ανασκευάσαμε διάφορους ισχυρισμούς, τα υπόλοιπα περιείχαν αναλύσεις στο μέτα επίπεδο και για το micro-targeting αλλά και για άλλα θέματα. Αυτό που διδαχτήκαμε από την προσπάθεια αυτή είναι εν τέλει ότι είναι σχετικά εύκολο να δείξει, να εξηγήσει κανείς σε πολλούς ανθρώπους σε σχετικά σύντομο διάστημα πώς λειτουργεί το fact-checking, να φτιάξουμε μια νέα ομάδα δηλαδή. Μάθαμε επίσης ότι είναι καλό να έχει κανείς στη διαθεσή του πολλά tools, πολλά εργαλεία, αλλά χρήσιμα είναι τελικά λίγα μόνο από αυτά είναι δύσκολο επίσης να παρακολουθούνται όλα. Αυτό που μάθαμε επίσης είναι ότι υπάρχει, είναι μεγάλη χρησιμότητα των communities. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε όλα όσα τρέχουν μέσα στα κοινωνικά ε, δίκτυα. Υπάρχουν και πολλά τα οποία κινούνται μόνο μέσα σε κλειστές ομάδες του διαδικτύου, μέσω WhatsApp και άλλων ε, εφαρμογών και για τα οποία ε, μας, επισημαίνουν, μας τα επισημαίνουν μόνο ενδιαφερόμενες κοινότητες. Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τα άρθρα μας τα δημοσιεύουμε, όπως είπα, μέσω του newsletter, αλλά και στα κοινωνικά μέσα. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να φτάσουμε και μέχρι τα άλλα μέσα, να τους ε, θα θέσουμε υπόψη δηλαδή, αλλά και τους multiplicators, έτσι ώστε να διοδοθούν τα άρθρα μας, τα οποία δεν διαδίδονται ακόμα μέσα στο διαδίκτυο. Αυτός ο δρόμος παραμένει κλειστός για εμάς μέχρι τώρα. Τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει είναι ιδίως ε, για θέματα μετανάστευσης και προσφυγικού και ε, προσώπων που ζητούν άσυλο, λιγότερο σε, άλλες, σε άλλους τομείς πολιτικής που έχουν φωτιστεί λιγότερο έως τώρα από την οπτική του fact-checking και εκεί κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια για παράδειγμα στον τομέα της υγείας. Δεν υπάρχουν και ιστοσελίδες fact-checking που να ανασκευάζουν συστηματικά ψευδείς ειδήσει. Τα περισσότερα fact, ε, τα περισσότερα ε, ε, fake news προωθούνται μέσω Facebook και κυρίως όταν πρόκειται για breaking news, δηλαδή για ε, τρομοκρατικές απόπειρες, για θεομηνίες καταστροφές κλπ. Εκεί παίζουν και τα social board καμιά φορά ένα ρόλο στην ενίσχυση το, της ε, διάδοσης των μηνυμάτων αυτών. Μέσω του Twitter, στη Γερμανία δεν υπάρχουν πολλοί χρήστες του Twitter, όμως μέσω του Twitter μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με, τους, με δημοσιογράφους. Όταν κάποιοι δηλαδή στέλνουν μέσω Twitter φωτογραφίες δίθεν εξαφανισμένων προσώπων και ούτω καθεξής, αυτά μετά τα παίρνουν τα, ε, τα, γνωστά μέσα και τα, τα, τα συνηθισμένα δηλαδή μέσα ενημέρωσης και τα διαδίδουν περαιτέρω. Fake news υπήρχαν στη Γερμανία και πριν αρχίσει η σχετική συζήτηση με την λεγόμενη κρίση του προσφυγικού ήδη από το καλοκαίρι του 2015 όταν κατέληξαν στη Γερμανία μεγάλες ε, ομάδες ε, προσφύγων και όπου άρχισαν να διαδίδονται πολλές ψευδείς ειδήσει σχετικά με τους πρόσφυγες αυτούς. Κάπω καθυστερημένα ήρθε και η αντίδραση των ε, μέσων ενημέρωσης αλλά και από την ε, πολιτική ελίτ σε ό,τι αφορά τι μεθόδους έχουμε πολύ λίγες ιστοσελίδες που ασχολούνται με fake news που διαδίδουν fake news Υπάρχουν όμως πολλά εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης τα οποία κάπου κάπου δημοσιεύουν και ψευδείς ειδήσει. Αλλά ασχολούνται και με άλλα θέματα ή ε, δημοσιεύουν πολύ επιλεκτικά κάποια πράγματα. Έχουμε κυρίως πολλές φωτογραφίες ή βίντεο τα οποία παρουσιάζονται εντελώς εκτός πλαισίου. Ένα παράδειγμα είναι πριν από τις εκλογές είχαμε ένα βίντεο που έδειχνε μια ομάδα 20 ανθρώπων περίπου σε, με λευκές φορεσιές που ε, περίμεναν σε μια στάση του μετρό στην Πιψία και αυτό ήταν δήθεν ο εξισλαμισμός της ε, Γερμανίας. Ψάξαμε και είδαμε ότι δεν ήταν οι άνθρωποι ε, μουσουλμάνοι, αλλά ήταν οι χριστιανοί από την Ερυθρέα. Ωστόσο το βίντεο αυτό το είχαν βγάλει από το πλαίσιο του και το δημοσίευαν ως ψευδός. Υπάρχουν και κάποιες επινοήσεις, ε, κάτι ε, ψευδείς δηλώσεις πολιτικών που διαδίδονται, φωτογραφίες, άλλα ντοκουμέντα. Αυτό που βρίσκουμε ότι λείπει ή πάντως θα μας βοηθούσε περισσότερο στην πράξη ήταν πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτό είναι το κλειδί για το λεγόμενο fact-checking. Δηλαδή από τις πλατφόρμες να έχουμε στη διάθεσή μας πολύ περισσότερα αριθμητικά στοιχεία, δηλαδή πόσα έχουν ε, δημοσιευθεί και διαδοθεί σε πόσους ανθρώπους έχουν φτάσει οι ψευδείς ειδήσει. Χρειάζεται μια συνειδητοποίηση και από πλευρά αρχών που πρέπει να αντιδρούν πολύ γρηγορότερα όταν για παράδειγμα η αστυνομία, οι αστυνομικές αρχές ή άλλες αρχές όταν αφορώνται αυτές είναι πολύ δύσκολο να έχει κανείς μια αντίδραση εκ μέρους τους αν δεν περιμένει πρώτα τρεις μέρες, αλλά μέχρι τότε έχει ξεπεραστεί, έχει κορυφωθεί η διάδοση της ψευδούς είδησης μέχρι να αντιδράσουν δηλαδή οι αρχές. Και βλέπουμε επίσης από την εμπειρία ότι όσο γρηγορότερα υπάρξει ανασκευή της δήλωσης, τόσο καλύτερα. Της ψευδούς δήλωσης εννοείται. Ειδικά για το ευρωπαϊκό πλαίσιο σημαντικό είναι επίσης να εξετάζονται τα συγκεκριμένα πλαίσια. Υπάρχουν περιφερειακές διαφορές. Υπάρχουν δίκτυα στη Γερμανία που παίζουν ε, σημαντικό ρόλο και γι' αυτό είναι σημαντική η δικτύωση και ανάμεσα στις ε, ιστοσελίδες που κάνουν το fact-checking. Και αυτό βεβαίως συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Κάτι που βρίσκουμε να λείπει ακόμη είναι να μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά και στις WhatsApp και στις κλειστές κοινότητες. Και ακόμη δεν έχουμε απολύτως καμία πρόσβαση σε, σε που κυκλοφορούν ανάμεσα στις ε, τουρκικές ε, κοινότητες και στις ρωσικές κοινότητες ε, στην Γερμανία που υπάρχουν πολλέ τέτοιε και εκεί βεβαίω εμεί δεν έχουμε καμιά απολύτω πρόσβαση στι ψευδεί ειδήσει που κυκλοφορούν σε αυτέ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ήταν αυτή μια πρακτική προσέγγιση στη δουλειά των fact-checkers που ελέγχουν τα στοιχεία που είναι πολύ σημαντική. και απαραίτητη δουλειά. Συχνά μιλάμε για αυτές τις, ε, τα δωμάτια με, την ηχό, την αντίχηση. Και το ηχείο, ε, κάπως έτσι λειτουργούν και εξαπλώνονται τα fake news. Βέβαια το θέμα είναι πώς θα μπει κανείς μέσα σε αυτή την αίθουσα τις ηχούς για να δει πώς ε, εξαπλώνονται οι ειδήσει πραγματικές και ψευδείς. Θα ήταν πολύ σημαντικό να δούμε ε, το τι παράγεται εκεί. Είναι και αυτή μια ε, σκέψη από την πλευρά μου. Λοιπόν, θα κάνουμε την ίδια διαδικασία. Θα αρχίσουμε με τους ε, συντονιστές και μετά θα δώσουμε το λόγο σε άλλους που θέλουν. Η Ζαμπίνε, μια ερώτηση έχω, σύντομη. Αν είχατε έναν ε, ε, εταίρο στο facebook στη Γερμανία, είπατε τέσσερις είναι δυνατόν να έχει κανείς αποτέλεσμα στον έλεγχο όταν έχει επιχειρήσεις όπως το Facebook που είναι πάρα πολλοί κόσμος εκεί ή μπορεί να γίνει έλεγχος χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα τεχνικά μέσα. Ε, να να είναι μόνο ε, ένα ποσοστό που να μπορεί κανείς να πιάσει ε, περιεχόμενα που να είναι σημαντικά για τους νέους ε, ή άλλες κατηγορίες. Σίλβια Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. σχετικά με τα όσα είπε ο καθηγητής κ. Δασκαλάκης, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, μάλλον να πω κάτι άλλο, το, να το πω διαφορετικά τα fake news ε, δεν είναι μονάχα το ίδιο το fake news, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως είδος ε, ως είδος που θα πρέπει να μπορούμε να το αναγνωρίσουμε ε, και ε, το οποίο κυρίως όταν συνδέεται με μια εσκεμμένη διαδικασία πρόθεσης. Εδώ θα μπορούσαμε επομένως να βρούμε αυτό που μερικοί μπορεί να πω να το ονομάσουν διαφάνεια και που εγώ το ονομάζω ευθύνη. Αναφερθήκατε στα ρομπότ ας πούμε, σε αυτά τα, τα οποία κάνουν κάνουν μία προώθηση εσκεμμένη και ενορχιστρωμένη. Επίσης δεν ξέρω πώς λειτουργεί ακριβώς ε, ε, αυτή η σχέση με το Facebook που έχει η άλλη ομιλήτρια, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχουν κάποιοι εταίροι, κάποιοι watchers, οι οποίοι θα παρακολουθούν αυτό το ε, κύκλωμα, γιατί αυτό το, αυτός ο κύκλος τώρα δεν είναι καθόλου ενάρετος, είναι φαύλος και επομένως θα πρέπει να το ξεπεράσουμε, να, βγούμε από τον φαύλο κύκλο, να δούμε πού ακριβώς και πότε ξεκινάει η ευθύνη το πρόβλημα όμως ε, ε, είναι ως εξής. Ε, όταν κερδίζουν χρήματα με το κάθε κλικ, όταν κερδίζουν χρήματα μέσα από τις διαφημίσεις, κανείς δεν πρόκειται να αποκαλύψει όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί πρόκειται πλέον και για στοιχεία τα οποία ενδεχομένως καλύπτονται και από το εμπορικό απόρριτο. Ερώτηση λοιπόν, λέτε κυρία Σφάτς, ότι έχουμε αυτή την εταιρική σχέση. Ε, κάνετε αυτές ε, τις ε, αναλύσεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες και κάνετε και κατάρτιση ακόμα πιο ενδιαφέρον. Όμως λέτε ότι από πλευράς του, του Facebook δεν μας απαντούν ποια είναι ακριβώς τα fake news. Δηλαδή στην ουσία δεν κόνουμε την ουρά μα. Πάμε γύρω γύρω. vielen herzlichen Dank, Herr Ευχαριστώ, κυρία Κατρούπ. Ευχαριστώ. Πριν από λίγες εβδομάδες είχα τη δυνατότητα να μιλήσω στον αρχή στην τάκτη του Euroactive τον Κρίστοφ Λεκλέρ και παραπονιόντουσαν για τα fake news. Δεν είναι καινούριο αυτό βέβαια στην ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά η διάδοση και η τεχνολογία τώρα διαφέρουν στην ψηφιακή επανάσταση. Και έλεγε ότι οι πλατφόρμες οι ψηφιακές δεν επενδύουν σε όλους αυτούς τους διορθωτικούς μηχανισμούς όπως το Corrective ή πολλές φορές πληρώνουν οι φορολογούμενοι για όλα αυτά και όχι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Γιατί αυτό δεν το δέχομαι, μας φορτώνουν με πολλά προβλήματα. Ε, αλλά πρέπει και εμείς να τους ε, βάλουμε ε, μπροστά στις ευθύνες τους. Ε, πώς χρηματοδοτούνται αυτές οι προσπάθειες και πώς ε, συμβάλλουν ε, οι εταιρείε σε αυτή την προσπάθεια ξεκαθαρίσματος και ε, αυτό ελέγχου. Ε, ε, ε, πάρα, πολλές, πάρα πολλοί φορείς ανήκουν στο Springer αλλά τα άρθρα τους είναι πραγματικά τόσο πολύ της μόδας και παρουσιάζουν την Μαργρέτα Φεστάγκερ ως μια παλιά σχολής κυρία. Ε, ευχαριστώ την εμπειρία με το πολίτικο την ε, είχαμε με τη μία ή την ε, άλλη μορφή και πραγματικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για έντιμη ε, δημοσιογραφία εδώ είναι στα όρια του fake news Μόρκανο δύο λεπτά Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και το πρώτο και το δεύτερο πάνελ εγώ θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα. Πρώτον, ε, εάν το πρόβλημα ήταν ε, απλό, δεν θα είμαστε εδώ τόσοι άνθρωποι να αφιερώνουμε χρόνο σε αυτό το ζήτημα. Ε, υπάρχει όμως, νομίζω, ένα πρόβλημα τώρα, το οποίο αφορά την επίγνωση της ποσότητας των πληροφοριών, των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά και των αρμοδιοτήτων. Και το λέω γιατί εμείς, σαν Επιτροπή Πολιτισμού, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το σκέλος της εκπαίδευσης γιατί πραγματικά εδώ πρέπει να δούμε ποιο είναι το περιεχόμενο, ποια είναι τα περιεχόμενα έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε συγκεκριμένες πραγματοποιήσιμες εφαρμόσιμες λύσεις. Δεύτερον, πάρα πολύ ε, ενδιαφέρον που ακούμε ότι για να σταματήσει λίγο αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει η τεχνολογία. Ξέρουμε πόσο γρήγορα αλλάζει η τεχνολογία. Επομένως το πρόβλημα είναι ποιος θέλει, ποιος έχει συμφέρον να αλλάξει η τεχνολογία έτσι ώστε να γίνουν πιο διαφανείς κάποιες διαδικασίες. Εάν δεν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα νομίζω ότι πάλι θα γυρνάμε γύρω-γύρω να δαγκώνουμε την ουρά μα. Ε, ε, ε, υπάρχουν αλγόριθμοι οι οποίοι βοηθούν την προώθηση ίσως θα μπορούσαν να βρεθούν και αυτοί οι αλγόριθμοι οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να μειωθεί σιγά σιγά η κυκλοφορία και η διάχυση. Ε, ε, ε, φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο μπορεί να βρεθεί τεχνολογικά. Αυτά είναι τα ζητήματα γύρω από τα οποία εμείς έτσι κάνουμε, προβληματιζόμαστε. Υπάρχει και κάτι άλλο όμως σήμερα είπαμε ότι έχουμε το Google, έχουμε το Facebook, ένα σωρό τέτοιες εταιρείες αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα sites τα οποία είναι στην ουσία σαν μια μαύρη τρύπα. Επομένως, τουλάχιστον στο όνομα της διαφάνειας είναι δυνατόν, τουλάχιστον λέω, ε, να, κάνουμε, να μπορούμε να κάνουμε μια επιτήρηση, ένα monitoring όσον αφορά την ιδιοκτησία ε, των sites Δηλαδή να ψάξουμε λίγο όχι μόνο τι είναι αυτό που φαίνεται εκ πρώτης όψεως αλλά να δούμε ποιος βρίσκεται από πίσω. Γιατί πίσω από μια, ένα κύκλο ψευδών ειδήσεων κάποιος ε, κρύβεται, κάποια συμφέροντα κρύβονται. Αυτά τα συμφέροντα πρέπει να αποκαλυφθούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ ο κύριος ε, βρήκα πολύ ενδιαφέρον και το δεύτερο μέρος και ιδιαίτερα την ε, ομιλία του συμπατριώτη μου, του κυρίου Δασκαλάκη, του καθηγητή Δασκαλάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ, γιατί είχε και λίγο αισιόδοξο τόνο. Δηλαδή ότι σιγά σιγά η τεχνολογία ενδέχεται να βοηθήσει, εάν βέβαια το επιθυμεί η πολιτική εξουσία, στην ε, θα έλεγα στη μείωση αυτού του φοβερού φαινομένου που είναι τα fake news. Και νομίζω ο συνάδελφος ε, Μόργανο τελευταία που μίλησε έθεσε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων αν μεταφράζεται αυτό ε, στο πώς και οι μεγάλες πλατφόρμες έχουν ειδική ευθύνη για αυτό το πράγμα και πρέπει να έχουμε και μια υπερηφάνεια στην Επιτροπή Πολιτισμού γιατί στο πρόσφατη έκθεση που ψηφίσαμε για τα πνευματικά δικαιώματα προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε λίγο το αυτό που λέμε καλό τύπο, τη δημοσιογραφία, αλλά και σε μια επόμενη έκθεση ε, για τα παράνομα κατά κάποιο τρόπο τις παρανομίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο πάλι η Επιτροπή Πολιτισμού θα καταβάλει νομίζω κάθε δυνατή προσπάθεια. Το συμπέρασμα είναι ότι το θέμα είναι πολύπλοκο αλλά αν τα αφήσει κανείς όσο πάει και θα γίνεται το τέρας θα αυξάνεται. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καιρός από πολλές κατευθύνσεις και η σημερινή νομίζω συνάντηση θα παίξει αυτό το ρόλο να φτάσουμε σε πιο πρακτικές αποφάσεις. Και έχω μια ερώτηση τελευταία προς τον κύριο Δασκαλάκη. Ε, εάν αυτό το φαινόμενο το fake news σιγά σιγά γίνεται και θέμα ερεύνης στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια που γνωρίζουμε ότι χρόνια τώρα πρωτοπορούν σε ερευνητικές διαδικασίες. Αυτό θα ευκολύνει τη λύση του προβλήματος, η καθαρά επιστημονική έρευνα. Ευχαριστώ πολύ. Σιόρτοβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις παρουσιάσεις και για το έργο σας πρωτίστως, για τις προσπάθειές σας. Μία ερώτηση στην κυρία Σουάρτς. Από ό,τι κατάλαβα, εργάζεστε σε μια οργάνωση μικρή. Έχετε και κάποιους εταίρους, δηλαδή δίκτυα, παρομοίων οργανώσεων, έχετε συνεργασίες. Και δεύτερη ερώτηση. Υποθέτω ότι θα έχετε και ιδιωτικές πηγές, αλλά έχετε και κάποιες δημόσιες ε, ε, πηγές χρηματοδότησης για να μπορείτε να συνεχίζετε το σημαντικό έργο σας. Ευχαριστώ κύριος ε, Μάλινος. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Λυπάμαι που έχασα την αρχή. Αλλά μέσα από τη συζήτηση ε, κατάλαβα αρκετά πράγματα. Θα είμαι ειλικρινής. Κι εγώ ήμουν ερευνητής, ε, πανεπιστημιακός, προσπάθησα να ασκήσω επιρροή. Ε, υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με την αρμοδιότητα, το χρόνο που δαπανάτε σε όλα αυτά τα θέματα. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε πάρα πολλές ε, ευθύνες και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη διατύπωσή μας. Πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, γιατί αυτό μπορεί να γυρίσει εναντίον μας ως πολιτικών. Για να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί και συγκεκριμένοι. Ε, απευθύνομαι εδώ στην κυρία Σουάρτς. Ας πούμε, ε, έχετε τέσσερις ανθρώπους στο γραφείο σας. Μπορείτε να δείτε το θέμα μέσα από το δικό μας πρίσμα. Αν είχατε πολιτική εξουσία, τι θα κάνατε. Πείτε μας λίγο γι' αυτό. Είναι πολύτιμο. Πιο πολύτιμο για μας από την ανάλυση που γίνεται. Να δούμε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Εμείς Έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο για να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατίες μας από παραβιάσεις, διαδικασιών, εξαγορά ψήφων κλπ. Αυτά έχουν περιγραφεί, έχουμε μαζέψει καλές πρακτικές, έχει ποινικοποιηθεί το θέμα κλπ. Γιατί, διότι έτσι ε, παραποιείται το εκλογικό αποτέλεσμα. Αν δεν έχουμε δίκαιες εκλογές, πώς θα έχουμε δημοκρατία. Ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Αυτό είναι η ελάχιστη προϋπόθεση. Και μετά μπορεί κανείς να προσθέσει και άλλα πολλά. Αν το δούμε μέσα από αυτό το πρίσμα, τα fake news, αν έχουν πολιτικά κίνητρα, είναι και το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει τώρα, ε, καταστρέφουν την ίδια τη βάση της ε, επιλογής του λαού. Δεν έχουμε ελεύθερε και δίκαιε εκλογές αν δεν ελέγχουμε τα fake news. Είναι ζήτημα χρόνου μέχρι να γίνει αυτό ευρύτερα κατανοητό. Είναι πάρα πολύ άδικο, όπως είναι άδικο να ε, ασκεί κανείς σωματική βία ή να εκβιάζει τους ψηφοφόρου όπως γινόταν στις αρχές του αιώνα. Έτσι λοιπόν σας καλώ πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις στο θέμα, θα πρέπει να πείτε ε, απευθείας στους πολιτικούς τι μπορούν να κάνουν, αν μπορούν, μέσα στο συνταγματικό τους πλαίσιο, το οποίο δεν είναι καθόλου έτοιμο για να μπορέσει να καταπολεμήσει τα fake news. Ευχαριστώ. μια γενική ερώτηση. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε οι πολιτικές πρωτοβουλίες να είναι αποτελεσματικές για τους πληθυσμούς, για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι λιγότερο εμπιστεύονται τους πολιτικούς και τα θεσμικά όργανα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Πώς μπορούμε να τους πιάσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Ευχαριστούμε πολύ και μία ή δύο ερωτήσεις από μένα την ίδια, αν μου επιτρέπετε. Μιλήσατε για αξιόπιστες πηγές. Όλοι εδώ θα μπορούσαμε, πιστεύω, σε λίγο διάστημα να συμφωνήσουμε τι σημαίνει για μας αξιόπιστες πηγές. Στην Γερμανία για πολύ καιρό ακούγαμε συχνά για τύπο ψευδών, τον τύπο δηλαδή που διαδίδει ψεύδι. Και αυτά από διάφορες πλευρές του πολιτικού φάσματος και που δεν αναγνωρίζουν πλέον έγκυρες ε, πηγές ε, ειδήσεων ως τέτοιες. Θα πούνε οι ίδιοι ότι δεν πρόκειται για αξιόπιστη πηγή. Και πρόκειται για ψεύδι, δηλώνουν αυτοί τα όσα διαδίδουν οι έγκυρες κατά τα άλλα εφημερίδες καθημάς δηλαδή. Η ερώτησή μου είναι για τον κύριο Δασκαλάκη. Αν κατάλαβα καλά τα όσα είπατε, μπορεί να μας βοηθήσει η τεχνολογία πολύ για να αποκαλύψουμε τις ψευδείς ειδήσει, τα fake news. Κάτι όμως πρέπει να ληφθεί πάντοτε υπόψη είναι όχι μονάχα η ίδια η καθεαυτό είδηση, πρέπει πάντοτε να δω και ποιο είναι το πλαίσιο με στο οποίο εμφανίζεται. Δηλαδή να κάνω μια παράλληλη ανάλυση τι άλλο έχει δημοσιευτεί για το ίδιο θέμα, από ποιε πηγές, αν υπάρχουν άλλες ειδήσει με όμοιο περιεχόμενο και αν αντιλαμβάνομαι σωστά όλα αυτά τα κάνουν ως τώρα αλγόριθμοι και ε, τεχνικά μέσα. Αλλά απέναντι σε αυτά οι αλγόριθμοι και τα τεχνικά μέσα είναι λίγο πολύ τυφλά. Επομένως δεν το είπα και τόσο αστειευόμενη ε, στην κυρία Σβάρτς ε, όταν της έδωσα το λόγο ότι χρειαζόμαστε και την ανθρώπινη παρέμβαση για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε την ψευδή είδηση. Χρειάζεται δηλαδή η παρέμβαση ενός ανθρώπου, ενός πραγματικού προσώπου που θα ελέγξει το περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκε η είδηση. Άρα θα πρέπει να ασχοληθούν πολύ περισσότεροι άνθρωποι με τα κοινωνικά μέσα ή να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες όπως αυτή της κυρίας Σβάρτς, γιατί αυτό που χρειάζεται είναι να αντιμετωπιστεί η μάζα των πληροφοριών που καταλήγουν στα ε, μηχανήματά μας ή στα τραπέζια μας. Να δώσω το λόγο όπως και πριν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά να κάνουμε με ένα τελευταίο γύρο εδώ με τους εμπειρογνώμονες του πάνελ. Ο κύριος Σαβίνη, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Ε, θέλω να υποβάλω ένα ερώτημα στην ουσία. Αυτό που προκύπτει από τα σχόλια και λοιπά είναι ότι το fact-checking είναι η άμεση απάντηση σε ένα νέο φαινόμενο. Ε, αλλά υπάρχουν και κάποια, ε, ε, κάποια κενά Ε, ίσως δεν έχουμε βρει ακόμα τα σωστά τεχνολογικά εργαλεία έτσι ώστε ε, να περάσουμε ε, στον έλεγχο των, όχι μόνο των προφανών ας πούμε fake news αλλά και των λίγο πιο περίπλοκων ε, επίσης ε, υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά την έλλειψη διασύνδεσης και μεταξύ κρατών και μεταξύ οργανισμών. Αυτά αποτελούν εμπόδια. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πρόβλημα, ίσως και μεγαλύτερο μάλιστα το οποίο προκύπτει. Δηλαδή πώς μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε τις, τα false news, τα fake news, τις ψεύτικες ειδήσει εν τη γενέση πριν αρχίζουν δηλαδή να ε, ε, προωθούνται και να διαχέονται. Ε, θα πρέπει η τεχνολογία να καθορίσει κάποια συστήματα όπου οι διάφορες παράμετροι, ε, ταυτοποίηση ε, πηγών, amplifiers που χρησιμοποιούνται, που μπορεί να είναι μηχανικά ή μπορεί να είναι άτομα, το στοχευμένο ακροατήριο κτλ. Μαζί με την ανάλυση του περιεχομένου, όλα αυτά μαζί να μπορέσουν να δώσουν μια απάντηση στο τι συμβαίνει στις διάφορες πλατφόρμες. Το Twitter δίνει κάποια πρόσβαση, άλλες πλατφόρμες δεν δίνουν καμία πρόσβαση τι είδους πρόσβαση στα δεδομένα θα πρέπει να έχουμε έτσι ώστε να έχουμε μια αξιοπρεπή, ε, ένα αξιοπρεπές tracking των ε, ε, ψευδών ειδήσεων. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες, θα πρέπει να καλωσορίσω και μια άλλη ομάδα επισκεπτών, μαθητές και μαθήτριες από τον Ντούσελντορφ, την πατρίδα μου. Καλώς ήρθατε λοιπόν και ελπίζω να αποκομίσετε κάποια πράγματα χρήσιμα από τη συζήτηση. Και τώρα θα δώσω... Ε, ναι, <laughs> αξίζει χειροκρότημα, ναι. Και τώρα Δίνω το λόγο στους δύο εμπειρογνώμονες. Δεν ξέρω ποιος θέλει να αρχίσει. Ε, μπορείτε να διαλέξετε ποιος αρχίζει πρώτος και ποιος θα απαντήσει σε ποιες ερωτήσεις. Έχω γράψει πολλά πράγματα. Θα τα πω γρήγορα. Για την κάμερα με την αντίχηση ε, και πώς μπορούμε να μπούμε μέσα εκεί. Υπάρχουν τεχνικές για να το κάνουμε αυτό. Ε, είναι εφικτό δηλαδή. Επίσης υπάρχουν τεχνικές λύσεις ε, με αλγορίθμους. Είχαμε αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας στο Las που δεν είχαν υπάρξει και αυτά είναι πολύ ψηλά στα αποτελέσματα στο Google και μετά προσαρμόστηκε ανάλογα ο αλγόριθμος για την αξιολόγηση και αυτό γίνεται. Για το Facebook και μέτρα ε, fact-checking έχουν γίνει κάποια, ε, κάποιες προσπάθειες. Όταν δηλωθεί κάτι ως λάθος ε, δήλωση, τότε υπάρχει 80% ε, λιγότερη αντίδραση, δηλαδή με like, tweet κλπ. Θα πρέπει όμως να περάσει χρόνος μέχρι να πάρουμε κάποια αποτελέσματα για διάφορους λόγους. Καμιά φορά η συνεργασία με τις αρχές καθυστερούν πρέπει να περιμένουμε πολύ μέχρι να απαντήσουν σε κάτι. Εμείς δεν είμαστε ομάδα που διαγράφει οτιδήποτε. Εμείς ε, τα παρακολουθούμε ε, ρητορική μίσους, εμπριστικά περιεχόμενα κλπ. Αυτά δεν μπορούμε να τα επηρεάσουμε. Για τους πόρους μας ε, ε, ελπίζομαι να ε, βελτιώσουμε τον οργανισμό, να ενταχθούμε και στην κοινότητα και να συνεργαζόμαστε και στο fact-checking με τοπικούς φορείς, ίσως και τοπικά μιμιέ. Καμιά φορά η εμπιστοσύνη απέναντι στα τοπικά ε, μιμιέ, ε, ε, η εμπιστοσύνη είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί υπάρχει μεγαλύτερη επαφή, μεγαλύτερη κατανόηση ε, σε τοπικό επίπεδο. Πολιτικά μέτρα δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κρατικές αρχές που θα λένε αυτό επιτρέπεται, αυτό όχι. Θα πρέπει να τάσσονται υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της δημοσιότητας, υπέρ της παρουσίασης στατιστικών δεδομένων, ε, σίγουρα χρειάζεται εκπαίδευση. Εκπαίδευση και για πιο μεγάλη ηλικίας ανθρώπους, γιατί ε, με τη δημογραφική εξέλιξη, στη Γερμανία τουλάχιστον, ε, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ψηφοφόροι επηρεάζουν τις εκλογές και εκείνοι χρειάζονται εκπαίδευση και σίγουρα ε, χρειάζονται πανευρωπαϊκά ε, επενδύσεις στην εκπαίδευση του δικαστικού και αστυνομικού σώματος. Σίγουρα ε, θα περάσει χρόνος μέχρι να γίνουν όλα αυτά, μέχρι να πιστούν για την ανάγκη. Τώρα, για τον τύπο του ψεύδους, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρω εδώ ένα πολύ καλό έργο που λέγεται Cyber Hate το οποίο καταγράφει σχόλια ε, σε ειδήσει. Ε, υπάρχουν πάρα, πολλές, ε, πάρα πολλά στατιστικά σχετικά με το πόσοι και ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τα περισσότερα σχόλια. μπορούμε να έχουμε ε, να παρακολουθήσουμε δηλαδή ε, τα σχόλια και τις πηγές τους και αυτό μπορούμε να το δούμε. Α, για τους, ε, τους οικονομικούς πόρους μας. Εμείς δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, ε, παίρνουμε από ιδρύματα και δωρεές, ιδιωτικά ιδρύματα και δωρεές ε, έχουμε οικονομικούς πόρους. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ακούστηκαν ορισμένα πολύ σοβαρά θέματα. Κράτησα κάποιες σημειώσεις, δεν μπορώ να τα καλύψω όλα αυτά που είπατε. Αρχίζω λοιπόν Ποιος έχει την ευθύνη των fake news για τα fake news. Αν τα, οι πλατφόρμες έχουν ευθύνη για τη διάδοσή τους. Όπως είπα, το fake news έχει ένα περιεχόμενο και όποιος γράφει το περιεχόμενο αυτό πρέπει να αναλάβει ευθύνη για το περιεχόμενο. Από την άλλη πλευρά, αν ένα άρθρο με fake news εξαπλώνεται γιατί πραγματικοί άνθρωποι το διαδίδουν, ενώ είναι ενορχιστρωμένη και κατασκευασμένη ε, καμπάνια από bots στο σκοτεινό δίκτυο ή ε, αν προωθείται από κυβερνήσεις. Οι πλατφόρμες ε, πρέπει να το σταματήσουν. Εάν κάτι παρουσιάζεται ως κοινωνικά ελκυστικό ενώ δεν είναι γιατί προωθείται μέσα από ενορχιστρωμένη εκστρατεία η ευθύνη είναι εκείνου που το παρουσιάζει ως κοινωνικά ελκυστικό. Και θα πρέπει να ε, κινηθούμε ώστε να εξαλειφθούν τέτοια φαινόμενα. για τα δεδομένα να πούμε μερικά πράγματα, γιατί τα δεδομένα είναι πραγματικό πρόβλημα. Όταν προειδοποιούμε για fake news, ε, μπαίνουμε σε θέματα ιδιωτικής σφαίρας των δεδομένων. Είναι δύσκολο οι fact-checkers που ελέγχουν τα δεδομένα δηλαδή να κάνουν τη δουλειά τους εδώ. Είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι ο fact-checker θα μπορεί να μπαίνει στα eco-chambers στους θαλάμους ε, αντίχησης και θα παρακολουθούν ε, τις ε, συζητήσεις που είναι ιδιωτικές. Από την άλλη πλευρά, οι αλγόριθμοι μπορούν να φιλτράρουν το περιεχόμενο. Οπότε, γιατί μιλάμε. Μιλάμε για συνομιλίες που γίνονται σε chat rooms. Εκεί είναι δύσκολο να γίνει παρακολούθηση χωρίς να παραβιαστεί η ιδιωτική σφαίρα. Αν από την άλλη μιλάμε για την διάδοση ενός άρθρου που έχει μια πηγή και έχει πάει, ανέβει κάπου στο ίντερνετ, το Google, το Facebook κλπ μπορούν να χρησιμοποιήσουν αλγορίθμους αλλά και ανθρώπους που ελέγχουν το, τα στοιχεία, τα πραγματικά. Με τα δεδομένα πρέπει να είμαστε πολύ ευαίσθητοι, γιατί και τα δεδομένα είναι ευαίσθητα και ιδιωτικά και πρέπει να τα προστατεύουμε. Οι αλγόριθμοι ε, δεν λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον ε, μέσα στο οποίο διαδίδονται τα fake news. Υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι. Υπάρχουν αλγόριθμοι που κοιτάζουν το περιεχόμενο, αλλά και αλγόριθμοι που βλέπουν τρόπους διάδοσης οι αλγόριθμοι γιατί ε, μια από τις μεγάλες ιδέες πίσω από το Google και τη μηχανή αναζήτησης είναι αυτό που μετράει δεν είναι τόσο το περιεχόμενο μια σελίδα, αλλά το πώς οι σελίδες διασυνδέονται. Η, διασύνδεση των περιεχομένων καμιά φορά είναι πιο σημαντική από το ίδιο το περιεχόμενο. Οι αλγόριθμοι το λαμβάνουν υπόψη τους αυτό. Είναι σημαντικό να λυθεί υπόψη. Και ανέφερα κάποιες ιδέες για το πώς μπορούν όλα αυτά να χρησιμοποιηθούν για να φτάσουμε στις πηγές και στο κίνητρο ε, διάδοσης fake news και να εντοπίσουμε τους τρόπους, τις μορφές διάδοσης. Ε, αν έχουν μπει στην έρευνα τα fake news, σίγουρα υπάρχει πολύ ενεργή έρευνα ε, δηλαδή η επεξεργασία φυσικής γλώσσας ε, για να επεξεργαστούμε το περιεχόμενο, αλλά υπάρχουν και αλγόριθμοι που προσπαθούν ε, να καθορίσουν μοτίβα συμπεριφοράς κλπ. Γίνεται επίσης δουλειά στην κατασκευή των bots, γιατί η τεχνολογία εδώ μας δίνει τρόπους να κάνουμε και καλά πράγματα και κακά. Ένας από τους ο της, της επιστήμης των υπολογιστών, ο Άλαν Τιούρινγκ, έγραψε ένα άρθρο για, στη δεκαετία του 50 για την τεχνητή νοημοσύνη και είπε ότι ε, αν το bot κάνει συζήτηση με έναν άνθρωπο χωρίς να τον πάρει είδηση ο άνθρωπος ότι είναι bot, ε, ε, τότε έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά όλα μπορεί να έχουν και αρνητικές επιπτώσεις. Ε, δεν ξέρω αν είδατε μια περίφημη υπόθεση πέρσι ή πρόπερσι όπου ένα πολύ καλό Twitter bot της Microsoft που ανέβηκε στο Twitter βρέθηκε σε ένα περιβάλλον ρητορικής μίσους και ρατσιστικών σχολείων και αλληλεπιδρώντας έγινε και το ίδιο ρατσιστικό. Δηλαδή το περιβάλλον το ανθρώπινο περιβάλλον μέσα στο οποίο βάζουμε την τεχνολογία, αυτό το περιβάλλον το ανθρώπινο αλλάζει και την τεχνολογία. Μπορεί να είναι καλές οι προθέσεις της τεχνολογίας, αλλά αν βρεθεί σε κακό περιβάλλον, ε, ε υιοθετεί προκαταλήψεις που, και λάθη του περιβάλλοντος. Ο έλεγχος των fake news λοιπόν είναι πολύ δύσκολη διαδικασία δεν θα μπορούσα να πω ότι θα μπορούσα να λύσω το πρόβλημα και είναι δύσκολο οι ρυθμιστικοί φορείς να προσαρμοστούν στις αλλαγές της τεχνολογίας επίσης. Τέλος, είναι σημαντικό ε, πρόβλημα στην έρευνα, είναι και ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με το διαδικτυακό γραμματισμό και την εκπαίδευση των χρηστών του διαδικτύου και σίγουρα το fact-checking, ο έλεγχος των ε, πραγματικών περιστατικών και οι φορείς που θα κάνουν αυτή τη δουλειά είναι πολύ σημαντικοί. Είναι όμως πολύ εργασιοβόρος αυτή η διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν αυτό. Οι αλγόριθμοι πρέπει να αναλάβουν μεγάλη από αυτή τη δουλειά. Και σε τελευταία ανάλυση υπάρχουν και φιλοσοφικές ε, συζητήσεις σχετικά με το τι είναι αλήθεια, τι είναι ε, fake κλπ. Και Τέλος, πιστεύω ότι πρέπει να προστατέψουμε, γιατί ο καθένας έχει μια φωνή, έχει λόγο και μπορεί να αρθρώσει λόγο στο βαθμό που δεν παραβιάζει ε, πολιτικά δικαιώματα, αλλά ε, εδώ παρουσιάζονται πράγματα όσοι αν διαδίδονται από ανθρώπους και οδηγούν σε εκστρατείες μεθοδευμένες. Αυτά πρέπει να περικόψουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα μπορούσαμε επί ώρες να συζητούμε το ίδιο θέμα. Βλέπω ότι ο κύριος Χέντριξ ζήτησε πάλι το λόγο. Να σας δώσω αμέσως το λόγο και να ολοκληρώσουμε. Με ρώτησαν για την άμεση πολιτική αντίδραση. Να σας πω λίγα πράγματα πολιτικοί φορείς, NGO, άλλοι φορείς που έχουν την ίδια ατζέντα όπως εσείς. Υπάρχουν πολλοί, ο ΩΣΑ, τα Ηνωμένα Έθνη, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Ζητήστε τους να συνδυάσετε τη δυνάμεις σας για να προκαλέσετε την αλλαγή. Νομοθετική ρύθμιση. Εάν κάτι σας φαίνεται ότι είναι τύπος, είναι τύπος. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχισυντάκτες τώρα είναι αυτοί που τρέχουν το Facebook, το Google και όλοι αυτοί και είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά που βγάζουν στις πλατφόρμες τους. Μπορείτε να ρωτήσετε πώς το κάνουν αυτό. Δεν είναι δικό σας το πρόβλημα αυτό των νομοθετών, είναι δικό τους πρόβλημα των αρχιστακτών. Μπορείτε να τα πείτε και σε όλους τους άλλους, από την Deutsche Zeitung, από το BBC και το Reuters. Μπορείτε να επιβάλλετε σε όλους αυτούς τα ίδια πρότυπα και δεν τα βάζετε και στο Google, Facebook κλπ. Τρίτο, βρείτε επιστήμονες για να συνεργαστείτε και να κάνετε την ε, γνώση και πάλι ελκυστική. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το Facebook για τις δικές σας δουλειές. Βρείτε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων που να έχετε κοινά συμφέροντα. Δεν είναι όλες κακές. Facebook και Google έχουν και αναλάβει πρωτοβουλίες για να καταπολεμήσουν τις κακές ειδήσει, τις, ε, τις ε, ψευδείς ειδήσει. Κάντε έρευνα και κάντε την τώρα δεν είναι και τόσο δύσκολο. Αυτά είχα να σας πω. Και το έβδομο, γιατί όχι. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος Κάμερ Έβερτ Αυτά με την ικανότητα χρήσης των ε, μέσων ενημέρωσης τα έχουμε συζητήσει και το πρωί. Πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη, να βοηθήσουν τους εαυτούς τους, γιατί δυστυχώς τα μέσα που διαθέτουμε είναι περιορισμένα. Όσο και να αγωνιζόμαστε ως Επιτροπή Πολιτισμού και να επιμένουμε και να πιέζουμε. Ευχαριστώ όλες και όλους τους εμπειρογνώμονες, δηλαδή τους εμπειρογνώμονες και την μοναδική εμπειρογνώμονά μας. Ήταν πραγματικά συναρπαστική η συζήτηση και πολύ ενημερωτική η σημερινή απογευματινή συνάντηση. Θα δούμε ποια συμπεράσματα θα μπορέσουμε να αντλήσουμε από την συζήτηση αυτή. Η συζήτηση θα συνεχιστεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στιγμή πιθανότατα μετά από τις σχετικές ακροάσεις θα υποβάλει κάποια πρόταση και θα επανέλθουμε ασφαλώς. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις παρεμβάσεις σας, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Εύχομαι καλό υπόλοιπο εδώ στις Βρυξέλλες, η, ε, η δεμή καλή επάνωδο στις αιστείες σας. Έχουμε ένα ακόμα θέμα στην ημερησία μας διάταξη και γι' αυτό παρακαλώ τα μέλη ευρωβουλευτές να παραμείνουν για λίγο ακόμη στην αίθουσα. Και βεβαίως δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα η συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Έχω λοιπόν να σας γνωστοποιήσω ότι το υπαριθμόν 11 θέμα της ημερησίας διατάξω συζήτηση για την έκθεση, για την εκτέλεση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την νεότητα, ότι αυτό το θέμα δεν μπορούμε να το συζητήσουμε σήμερα, διότι η συγγήτρια είναι δυστυχώς ασθενής και κολλείεται να προσέλθει αλλά δεν μπορούμε και να το αναβάλουμε για φέτος. Άρα θα μπούμε αμέσως με τον Ιανουάριο, αμέσως τον Ιανουάριο μάλλον, στην υποβολή της εκθέσεως και στη συζήτησή της και την ανταλλαγή απόψεων, η οποία προβλεπόταν σήμερα όπως σας εξήγησα. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να αναβάλουμε, είναι δυστυχώ ασθενή η συγκίτρια δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Μα μένει ένα τελευταίο θέμα τη ημερησία διατάξεως, για το οποίο θα παρακαλέσω όλοι να εγκαταλείψουν την αίθουσα, όσοι δεν ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό βεβαίως ισχύει, που λέω, και για τους συνεργάτε και συνεργάτηδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι στην αίθουσα θα παραμείνουν μόνον ευρωβουλευτές και συνεργάτες τους αυτών και των πολιτικών ομάδων.